Dear colleagues, I'm going to... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσω τη συνεδρίαση εγκαίρως, στην ώρα μας. Θα κάνω τις ανακοινώσεις του Προέδρου και μετά θα συνεχίσω Αφήνοντα ένα μικρό διάλειμμα πριν από την ψηφοφορία. Από ό,τι κατάλαβα προσέρχονται σιγά σιγά οι συνάδελφοι. Θα ήθελα πάντω να αρχίσω με τις ανακοινώσεις. Πριν από την ψηφοφορία θα ε, επιβεβαιώσω ότι είστε όλοι παρόντες. Να κάνω λοιπόν τις ανακοινώσει του Προέδρου τώρα. Καταρχά, θα ήθελα να σα πω ότι θα γίνουν οι εξή αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη οι συντονιστές αν μ' ακούνε θα είναι χρήσιμο αυτό για το 18, το EU Lisa. Θα γίνει στις 10 και 4 αντί στις 10.45. Παρακαλώ οι συντονιστές τουλάχιστον να με ακούτε. 18 για το EU Lisa θα λάβει χώρα στις 10 και 4 αντί για 10 και 45. Επίσης προστίθεται το σχέδιο έκθεσης για την ε, στρατηγική ψηφιακού εμπορίου στις 10 και 45. 10, 11, 12 για το πακέτο SAS έχουν αναβληθεί ε, για τις 16 Νοεμβρίου όσον αφορά το 18 για την νομιμοποίηση ε, προσόδων από, από, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε, το 20 για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα ΕΦΗ, e e συστήματα μεταφορών έχει ε, ακυρωθεί. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορεί μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν θα υπάρχει διερμηνία από τα κροατικά και τα γαλλικά. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη είναι η συγγήτρια για το, την έκθεση πρωτοβουλίας ε, για την ελευθερία των, και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Ο Κώστας Δεσκόνης ε, ε, για τη γνωμοδότηση των απαλλαγών για το 2016 για την Europol, τη Eurojust, τη Frontex, το FRA όπως επίσης και για τις εκθέσεις, τις οριζόντιες εκθέσεις των υπηρεσιών. Υπάρχει επίσης και το χρονοδιάγραμμα για τις επιτροπές ε, και τις συνεδριάσεις του 2018. Στις 12 Οκτωβρίου έλαβε ένα σχέδιο απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι μια ε, εκτελεστική πράξη για το 2020, κάτι το οποίο το λάβατε όλοι φαντάζομαι μέσω του newsletter Επιτροπολογία. Υπάρχει και μια εσωτερική προθεσμία για ε, ενδεχόμενες αντιρρήσεις, παρακαλώ ενημερώστε μας πριν από τις 27 Οκτωβρίου του 2017. Και όπως γνωρίζετε ε, θα γίνει σήμερα 8 η ώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να επιβεβαιώσετε ότι έχετε μαζί σας την κάρτα ψηφοφορίας γιατί θα ψηφίσουμε τα πάντα ηλεκτρονικώς. Συνάδελφοι, μπορείτε παρακαλώ να κάνετε μια σχετική ησυχία. Δεν θα αρχίσει η ψηφοφορία αν δεν ελέγξω με τους συντονιστές ότι είστε όλοι έτοιμοι. Μην ανησυχείτε λοιπόν, αλλά καθίστε παρακαλώ. Κυρία Βίξτρομ, έχετε το λόγο διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάρω το λόγο για λίγο. Δεν κάνουμε την ψηφοφορία ακόμα, κυρία Βίξτρομ. Θα κάνουμε ενό λεπτού συγγύη για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου. Παρακαλώ καθίστε. Δεν θα αρχίσουμε αν δεν είστε όλοι έτοιμοι. Λίγο την προσοχή σας θα ήθελα παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Μην μιλάτε λίγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως θα γνωρίζετε, στις 16 Οκτωβρίου η Δάφνη Καράνη διευρυνητική ε, δημοσιογράφος δολοφονήθηκε. Μπορούμε παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή και παρακαλώ όσοι προσέρχεστε ησυχία. Η Δάφνη Καράνα Καλίτσια γνωρίζετε πολύ καλά ότι δολοφονήθηκε ε, εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως Επιτροπή, γιατί μας ε, απασχολούν όλος ιδιαίτερος τέτοιου είδους σημαντικά ζητήματα. Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος ήταν πάρα πολύ ενεργός ε, στην ενημέρωση ε, ορισμένων των πολιτών για πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως τα έγγραφα του Παναμά. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω ενός λεπτού σιγή. Παρακαλώ πολύ. Thank you very much, Collins. Ευχαριστώ πολύ. So, colleagues, we now... Συνάδελφοι, περάσουμε λοιπόν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να αρχίσουμε με την ψηφοφορία του Δουβλίνου. Η κυρία Βίξτρομ θέλει να πάρει το λόγο πριν αρχίσουμε την ε, ψηφοφορία. Θα ήθελα να ελέγξω όμως, να εξασφαλίσετε, να επιβεβαιώσετε ότι όλοι είναι παρόντες ε, και να με ενημερώσετε αν ε, δεν ισχύει αυτό. Κυρία Βίξτρομ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ήταν πολύ μακρύ το ταξίδι μας μέχρι τη σημερινή ψηφοφορία και σήμερα έχουμε και δύσκολη μέρα μπροστά μας. Θα ήθελα να ε, σας ε, ευχαριστήσω επί τη ευκαιρία όλους, πραγματικά ολόκαρδα ε, προς όλη την ομάδα που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, χωρίς την αφοσίωση, την υπομονή των σκιωδών εισηγητών και των ομάδων τους και, την, συναδέλφους στην υπηρεσία μας, στην υπηρεσία την νομική και στην, ε, στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα. 21 συναντήσεις και οδόν εισηγιστών ε, ε, ποτέ δεν έχουν γίνει τόσες πολλές ε, συνεδριάσεις σκιωδών, πάρα πολλές τεχνικές συνεδριάσεις και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που προσπάθησαν οι συνάδελφοι να καταλάβουν ε, τις απόψεις όλων των άλλων συναδέλφων προσπαθώντας να διατηρήσουν την υποστήριξη των δικών τους ομάδων. Έδισαν λοιπόν την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί σήμερα να μιλήσει με μια ενωμένη φωνή που είναι κατά κάποιο τρόπο και ιστορική και μπορεί επίσης να αποτελέσει έμπνευση για το Συμβούλιο και τις σχετικές διαπραγματεύσεις και στους διαπραγματευτές μας βεβαίως. Σε σχέση βέβαια με αυτό που είπαν ε, στο Ευρωβαρόμετρο οι Ευρωπαίοι πολίτες, 70% είπαν ότι θέλουν η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το θέμα της μετανάστευσης. Αυτό λοιπόν είναι ο ακρογωνιαίος λήθος μας θέλουμε να δούμε μια ρεαλιστική προσέγγιση του ε, συστήματος ασύλου, του ευρωπαϊκού, που θα είναι δίκαιη και θα ακολουθεί τις βέλτιγες πρακτικές. Ελπίζουμε ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα ευρώ σήμερα και ότι το Συμβούλιο μπορεί να εμπνευστεί από το πνεύμα πραγματισμού ε, και συνεργασίας που οδήγησε το Κοινοβούλιο μας ε, στη σημερινή ψηφοφορία σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλους και ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βίξτρομ. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Κύριε Τσεδόφσκι, θέλετε κάτι να πείτε. Γιατί δεν υπάρχει ε, διερμηνία στα τσεχικά. Ε, πάρα πολλοί συνάδελφοι θα θέλαν ε, να ακούσουν σήμερα και πάρα πολλοί στο διαδίκτυο θέλουν να ακούσουν στα τσεχικά τι ακριβώς θα γίνει εδώ σήμερα. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εγώ έχω στείλει στον πρόεδρο το αίτημά μου για διερμηνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Θα δούμε για ποιο λόγο δεν υπάρχει διερμηνία. Ε, τσεχική σήμερα, ειδικότερα στη σημερινή συνεδρίαση που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη και στους τσέχους συναδέλφους σας. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει μου λένε εδώ οι συνάδελφοι. Υπάρχει τσεχική καμπίνα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε με την ψηφοφορία και θα το ελέγξω. Ας περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Έχω μια τεχνική ε, ανακοίνωση. Ακούστε με προσεκτικά. Για, τα άρθ, για το άρθρο 42 παράγραφος 1 υπάρχει ένα πρόβλημα τροπολογία 965 θα έπρεπε να λέει ότι καταπίπτει. Εάν η 961 μέχρι η 965 ή οι 8 εγκριθούν. Ας περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία και αρχίζουμε με την τροπολογία 110, 111, 112 που είναι ταυτόσιμες. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. closed. Πέρας. That is rejected. Απορρίπτεται. Κύριε Σπινέλη, δεν έχετε την κάρτα σας, δεν δουλεύει. Είναι σημαντικό να ψηφίσετε όλοι. Μήπως θέλετε να αλλάξετε, να αλλάξετε θέση και να βάλετε την κάρτα σας ε, σε ένα άλλο μηχάνημα. Μήπως εκεί δουλεύει. Συνάδελφοι, θέλω να είμαι βέβαιος ότι όλοι σήμερα θα ψηφίσετε. Άρθρο 2, συμβιβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Άρθρο 1, τροπολογία 286-287. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Συμβαστική 2 έναρξη ψηφοφορίας. Συγγνώμη, συγγνώμη, τροπολογία 300 έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα συμβιβαστική 2. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Έναρξη ψηφοφορίας. σελίδα 17 βρίσκεται. Συμβιβαστική 3 επαναλαμβάνω. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Έναρξη ψηφοφορία. Σελίδα 19. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Σελίδα 32. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Σελίδα 40. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9, σελίδα 41, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10, σελίδα 44, έναρξη. Πέρασε εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11, σελίδα 45, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12, στην ίδια σελίδα 45. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13, σελίδα 46, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14, σελίδα 48, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15, στην ίδια σελίδα 48, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16, σελίδα 49. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17, σελίδα 49. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασα. Γκρίνεται. Συμβιβαστική 18 σελίδα, 51, ε, συγγνώμη, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19, σελίδα 53, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Σελίδα 54, έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21, σελίδα 55, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 σελίδα 57. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 σελίδα 58. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 24, σελίδα 59, έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Άρθρο 25, 697, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25. Σελίδα 60. Έναρξη ψηφοφορίας. «702 Α, συγγνώμη, συγγνώμη, πέρα τη ψηφοφορία ξέχασα να το πω. Εγκρίνεται. Λοιπόν, είδατε πόσο δεδομένα τα παίρνω. Okay. 720 701, 702 είναι ταυτόσημες. Σελίδα 61, έναρξη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 26, σελίδα 63, έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27, σελίδα 67. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 769. Έναρξη ψηφοφορίας. Ναι. 769. Σελίδα 70. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 86. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94, 871 και 872 και η 873 μέχρι, τις την 880, σελίδες 83 και 84. Όλες αυτές είναι ταυτόσισμες. Έναρξη ψηφοφορίας. Το καταλάβατε? Mm. Λοιπόν, 94 μέχρι 880 τροπολογίες. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική 31, σελίδα 89. Συμβιβαστική 31. Έναξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32 σελίδα 90. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 953, 954, 955 και 956 σελίδα 93 αυτές ψηφίζουμε τώρα. Έναρξη ψηφοφορίας. Συνάδελφοι, λάθος μου. Ακυρώνουμε αυτή την ψηφοφορία. Πρώτα τη συμβιβαστική 33 πρέπει να ψηφίσουμε. Στη σελίδα 92 πάνω πάνω. Συγγνώμη, δεν την είδα. Συμβιβαστική 33. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Τη συμβαστική 33. Πέρας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. Τώρα πάμε στην 953, 954, 955, 956 ταυτόσημε σελίδα 93. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Κυρία Στίβενς, Μπορώ να κλείσω αυτή την ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, κυρία Στίβενς. Συγγνώμη, Πρόεδρε, που σας διακόπτω. Όμως, πάντα μας λέτε τον αριθμό της σελίδας, όμως αυτό αφορά μόνο τους καταλόγους ψηφοφοριών της δικής σας ε, ομάδας. Να μην λέτε λοιπόν ε, τις, ε, τους αριθμούς των σελίδων, γιατί εμείς έχουμε τελείως διαφορετικά στοιχεία. Να λέτε λοιπόν τις συμβαστικές, αλλά όχι τις σελίδες. Ευχαριστώ. Okay. Ναι, είναι ο κατάλογος που έχω του Προέδρου, δεν είναι ο κατάλογος των Σοσιαλδημοκρατών, όχι, εντάξει. Δεν θα αναφέρω τον αριθμό των σελίδων, θα αναφέρω μόνο τους αριθμούς των τροπολογιών. Συγγνώμη. 9.57. Άρχεται ψηφοφορία. Περάς. Απορρίπτεται. 9.58. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 97. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 9.60 έως 9.64 ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 98. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ενέξτε εννέα έως 9.74 ταυτόσιμες έρχεται. Πέρας. Έγκρινε. Συμβαστική 34. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. Συμβαστική 35. Έναρξη. Πέρας. Έγκρινεται. Συμβαστική 36. Έναρξη. Πέρας. Έγκρινεται. 9.91. Έναρξη. Εννέα, Πέρας. Έγκρινεται. Άφετ 23. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. 93. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 94. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 9, 96. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 9, 7. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 37. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38. Εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. Δέκα, έντεκα. Έναρξε. Δεν λέω αριθμό σελίδε, έτσι. Βλέπετε. Δεν το ξανακάνω αυτό το λάθο. Λοιπόν, τροπολογία 10-11. 1011. Ψηφίσατε, πέρας. Απορρίπτεται. 108 και 1012 αυτός μας άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 113. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 114. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 115. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 116. Έναξη. Πέρας. Αγκρίνεται. Τελογικές σκέψεις. 118. Πέρας. Απορρίπτεται. 119-120 μας άρχιδε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 123. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. ΑΦΕΤ 2. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 137. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Αφετ 7. Θα σας αφήνω να βρείτε μόνο στη σελίδα. Εγώ δεν σας τη λέω πάντως. Εγώ ψήφισα. λογική σκέψη 26, να σας δώσω ένα στοιχείο. Κυρία Γκόμες, δεν τη λέω τη σελίδα. Δεν επιτρέπεται. Συνεχίζει η ψηφοφορία, δεν ξέρω αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας, εγκρίνεται. 265. εξήντα πέντε. Ετολογική σκέψη 38. 265 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 268. Έναρξη. Απορρίπτεται. Αφέτ εννέα. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 269. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.77. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση επί του κειμένου όσο έχει τροποποιηθεί, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 43 ψήφοι υπέρ 16 κατά καμία αποχή. Τώρα επί της απόφασης ε, να μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 41 ψήφους υπέρ, 14 κατά. Σε χαρητήρια στην κυρία Βίξτρο. Καλή επιτυχία. Thank you so much and sorry for my mistake. Thank you colleagues for your discipline in that voting session. Very... Ευχαριστούμε για την επιθαρχία. colleagues, we do need to move um, promptly to the next. Uh, Πρέπει να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία, ταχύτατα. Συγχαρητήρια σε όσους ενδιαφερόμενους της πρώτης ψηφοφορίας. Προχωράμε τώρα. Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδείας Ταξιδίου Αίτιας. Εισηγήτρια κυρία Κίνγκα Γκάιλ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης, συμβούλους, βοηθούς και τη γραμματεία Νιγκάθρινη για όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Εκτιμώ ιδιαίτερως λοιπόν τη συνεργασία μας. Παρότι δεν συμφωνούσαμε σε όλα, νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και ελπίζω αυτό να φανεί και στις ψηφοφορίες. Thank you very much uh, to Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Συμβαστική για το άρθρο 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν ακούσαμε καλά, γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν τον κατάλληλο ψηφοφορία, να ξέρετε. Μπορεί να ήταν και 70. Συνάδελφοι, να εξηγήσω. Ησυχία, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε ψηφορία σε κατά τμήματα. Η διαδικασία Β είναι πρώτη. Και μετά θα ψηφίσουμε επί της τελικής έκθεσης. Συμφωνείτε? Ωραία. 70 και 82 λοιπόν συμβαστική και μετά περνάμε στις τελικές ψηφοφορίες. Στο άρθρο 70 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική λοιπόν τροπολογία για το άρθρο 70. Διαδικασία πριν από την τελική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 82. Άρχεται. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε λοιπόν από το κειμένο όσο έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση. Άρχεται. 42 ψήφοι υπέρ, 13 κατά και 3 αποχές. Επί της απόφασης τώρα να μπούμε σε διαπραγματεύσεις, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 43 υπέρ, 13 κατά, μία αποχή, σε την συγκήτρια. Πάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα. Η κύρια, κύριος κατάλληλος προφοριών που έχετε, 146, 147, 148, ταυτόσιμες έρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Εντάξει, είμαστε όλοι Okay. Ε, άρχεται η ψηφορία. Συμβαστική 1. Πέρας. γίνεται. 3.37 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Σημαντική στο άρθρο 2. Άρχεται. Πέρασε. Αγγλίνεται. Συμβαστική του άρθρου 3. Άρχεται. αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 4 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 6 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.90. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική στο άρθρο 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 8 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 9 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 10 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 10α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεβαστική του άρθρου 13. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Σεμβαστική στο άρθρο 14. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Για τη διαγραφή της παιδείας. Ομοδική ψηφορία. Εάν έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά για τη διαγραφή του occupation, έναρξη. Πέρασμα. Εγκρίνεται. Για τη διαγραφή του IP address, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Έναρξη. Πέρας. Έγινε Έγινε ναι. Πέντε δώδεκα, τροπολογία, πέντε δώδεκα, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Σεβαστική 16. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεβαστική στο άρθρο 17. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 19. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 20. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σημαστική του άρθρου 21. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεβαστική του άρθρου 22. Έναρξη. Πέρασε. Έγκρινεται. Σεβαστική το άνθρωπο 23. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτα τέσσερα έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Έναρξη. Πέρας. Εκρίνεται. Σεβαστική στα άρθρα 26 και 26α. Έναρξη. Πέρασε. Συνάδελφοι, ορισμένοι από εσάς δεν ψηφίζετε. Αν δεν θέλετε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, πέρασε. Ξέρω ότι είναι κουραστικό, αλλά να ψηφίζετε παρακαλώ. Έγκρινεται. Στο άρθρο 27. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 28, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο άρθρο 29 και 29α. Έναρξη. Πέρας. 758 έναρξη. Πέρασε. Απορρίπτεται. Στάθο 30, συμβαστική άρχεται. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Συμβαστική του άρθρου 31. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τριάντα δύο. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τριάντα τρία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική το 34. Φαίνεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεβαστική το 35. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Έναρξη. εγκρίνεται. 37 έναρξη. Πέρα. Εγκρίνεται. 38 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 8.75. Ε, ναι. Πέρα. Απορρίπτεται. Σεβαστικής άρθρο 40. Άρχεται. Πέρας. Γκρίνεται. 41. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 42. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεβαστική στο άρθρο 43. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Άρχεται. Εγκρίνεται. 45 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 47 άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. 48. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο 49. Άρχεται. Πέρας. Στο 50 τώρα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 52. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 52α. Άρχεται. Εγκρίνεται. 53. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική στο 54. 53α μάλλον. Πέρας. Εγκρίνεται. 54. Άρχεται. Πέρας. 55. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 56. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. 58 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 59 άρχεται. Πεντανέα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 60. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 62. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 63. Έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 64. Έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 65. έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 66. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 67. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 69. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 1037, 1037, άρχεται. Απορρίπτεται. Συμβαστική στο άρθρο 72, άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 73, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. τέσσερα. άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 75 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 76 έναρξη. Δεν Εγκρίνεται. 77 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 78 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 81 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ονταδύο σε παράρτημα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρχεται ψηφορία λοιπόν επί των ε, citations και recitals. σφαίρα, εγκρίνεται τροπολογία 163. Δεν σας τη λέω τη σελίδα, ό,τι και να λέτε. 163. Βρείτε τη σιγά σιγά. Τη βρήκατε. Μα είναι ανοιχτή η ψηφοφορία μέχρι να τη βρείτε. 163. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 177. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε να ψηφίσουμε το κείμενο έχει τροποποιηθεί μας έχει κλίση. Άρχεται. Πέρασε. Έγκρινεται με 42 ψήφους υπέρ, 12 κατά, 2 εποχές. Τώρα για την απόφαση ε, διαπραγματεύσεων άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται με 39 υπέρ, 13 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Um, Καθήστε, καθίστε, μη φεύγετε, για να κάνω μια τελική ψηφοφορία στην ε, έκθεση της κυρίας Χιμένεθ. Τερέσα Χιμένεθ Μπεθερίλ Μπάριο. Για τα ναρκωτικά. Συνεχίζουμε την ψηφοφορία είναι απόφαση πλαίσιο για τις ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Τερέζα, θες να πάρεις το λόγο πριν ξεκινήσουμε. Παρακαλώ ησυχία συνάδελφοι, να κάνουμε αυτή την τελική ψηφοφορία. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. Πάμε στο κείμενο αυτό. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 50 ψήφοι υπέρ, 4, κατά, 4 ψήφοι κατά, καμία αποχή, συγχαρητήρια. Κυρία Χιμένεθ Μπεθερίλ. Dear colleagues, συνάδελφοι, πάμε στο σημείο 7. Όλοι πιέζεστε χρονικά. Καλό θα να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καθίστε, εάν σας ενδιαφέρει να ακούσετε αυτό το σημείο. Το σημείο 7 είναι η παρουσίαση από τον Επίτροπο King του πακέτου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που υιοθετήθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων στις 18 Οκτωβρίου. Θα έχετε δει την ε, παρουσίαση πολλοί από εσά. Το πακέτο που παρουσιάστηκε χθες έχει μέτρα για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη για την προστασία του δημοσίου χώρου, καθώς και μέτρα για να μειωθεί η πρόσβαση στα μέσα που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, επικίνδυνες ουσίες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Είχε καλή υποδοχή αυτό το πακέτο χθε, έγινε ανάλυση επίσης τη πρόταση. Σήμερα όμως έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε ε, την παρουσίαση του Επιτρόπου μαζί με τον Επίτροπο. Έχουμε και συναδέλφου από τη νέα Επιτροπή που ασχολείται με την τρομοκρατία και, την, ε, και η πρόεδρος, ε, η κυρία Γκρίνσπεκ, είναι επίσης μέλος και της δικής μας Επιτροπής και Διάφορα άλλα μέλη είναι παρόντα από την Επιτροπή αυτή, τη Νέα Επιτροπή για την Δημοκρατία. Πολύ ωραία. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Επιτροπή, που σας έχουμε εδώ για να μιλήσουμε για την παρουσίαση αυτή. Το άλλο βασικό σημείο είναι να ακούσουμε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά για το PNR. Στις 26 Ιουλίου το ε, Συμβούλιο είπε ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδάς για το PNR δεν θα ολοκληρώνονταν στην, στην πρόσφατη μορφή, γιατί υπήρχαν ε, ασυμβατότητες με τα θεμελιώδη δικαιώματα της χάρτας. Ε, στις 7 Σεπτεμβρίου ακολουθήσαμε την, ε, το θέμα, γράψαμε ε, στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο ε, με απόψεις για τις επιπτώσεις της απόφασης. Για αυτά τα δύο βασικά σημεία θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο για μια παρουσίαση. Έχουμε πίεση χρόνου. Έχουμε μέχρι τις 10, γύρω στις 10 ας πούμε για αυτό το θέμα. Θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις, ε, πολύ σημαντικές ερωτήσεις ε, από ανθρώπους που ξέρουν. Α, είναι και η πρέσβη εδώ, συγγνώμη. Θα ακούσουμε και από την πρέσβη. Καλώς ήρθατε λοιπόν κι εσείς. Θα ακούσουμε και από την πρέσβη την άποψη την άποψή της δηλαδή. Καταρχάς θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο. Παρακαλώ να κάνετε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό να έρθω το συντομότερο δυνατόν εδώ στο Κοινοβούλιο για να κάνω μια ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα αυτά που πέρασε το Σώμα των Επιτρόπων χθε. Που υιοθέτησε το Σώμα των Επιτρόπων χθε. Σας ευχαριστώ που καταφέραμε σήμερα το πρωί να το κάνουμε αυτό. Θα χρειαστώ να φύγω, ζητώ συγγνώμη, λίγο μετά τις 10, γιατί θα πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο για να πάω στη συνεδρίαση G7, όπου θα συναντηθούμε και με την προσωπία την Αμερικανική και την Καναδέζικη. Όπως είπατε, τα μέτρα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο έχουν σαν σκοπό να αυξήσουν την ανθεκτικότητά μας, να έχει μικρότερη πρόσβαση να έχουν οι τρομοκράτες ε, στα μέσα που χρησιμοποιούν και να υπάρξει διεθνή συνεργασία. Ε, στα μέτρα που παίρνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως το τελευταίο χρόνο, αλλά να διδαχθούμε και από τις τρομερές ε, επιθέσεις του καλοκαιριού, οι οποίες έδειξαν ακόμα ότι η τρομοκρατική απειλή είναι πολύ πραγματική και συνεχής. Το είπα και το ξαναλέω. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε όλες τις επιθέσεις, δεν μπορούμε το υποσχεθούμε αυτό, δεν υπάρχει δυναμικός κίνδυνο, αλλά προοδευτικά μπορούμε να μειώσουμε τα παραθυράκια και τις πόρτες μέσα από τις οποίες περνάνε τρομοκράτε και λειτουργούν και μπορούμε να ανταποκριθούμε και να προσαρμοστούμε κι εμείς καθώ εκείνοι αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν, το ε, βλέπουμε ότι περνάμε σε μια τεχνολογία ε, χαμηλής τεχνολογίας. Ε, ε, ξεκίνησε την Νίκαια, ε, Βερολίνο, Στοκχόλμη, Βαρκελόνη κτλ. Λοιπόν, αντιγράφτηκε μετά δηλαδή στις άλλες πόλεις. Ε, με τη βοήθεια του ISIS ε, οι τρομοκράτες ε, πλήττουν ε, δημόσιες ε, συγκεντρώσεις, δημόσιες ε, πλατείες, αεροδρόμια, εκεί όπου συγκεντρωνόμαστε κτλ. Συγκεντρώθηκα, πριν από λίγες εβδομάδες συναντηθήκαμε με 60 δημάρχους στην Νίκαια και σε μια δήλωση οι δήμαρχοι ζήτησαν να καταρρεθούν περισσότερες προσπάθειες για να προστατευτούν οι δημόσιοι χώροι. Χθε λοιπόν ξεκινήσαμε ένα σχέδιο δράση, ούτω ώστε οι δημόσιοι χώροι να είναι λιγότερο ευάλωτοι. Χωρί χωρίς να αλλάζουμε όμω το βασικό, βασικά ανοιχτό χαρακτήρα τη κοινωνία μα. Υπάρχουν διάφορε λύσει. Κάποιε είναι φυσικέ ε, με εμπόδια, ε, τροχοπέδε, ε, που είναι και αυτέ χαμηλή τεχνολογία, αλλά το να τι εγκαταστήσουμε αυτές τις, αυτά τα μέσα να τα εγκαταστήσουμε είναι τα πανηρά. και οι δήμοι και οι κοινότητες μας λένε ότι θέλουν βοήθεια για να γίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, βρήκαμε 18,5 εκατομμύρια ευρώ για φέτος από την ε, χρηματοδότηση για την ασφάλεια και μέχρι 100 εκατομμύρια για του χρόνου ε, από τα περιφερειακά ταμεία ε, για τις καινοτόμες αστικές δράσεις. Υπάρχει και ένα φόρουμ για την διαφορετική συνεργασία επίσης για να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές ανάμεσα στις διάφορες αρχές και για να υπάρξουν δεσμοί ανάμεσα στις δημόσιες αρχές και στον ιδιωτικό τομέα τμήμα της ε, μεγαλύτερης προσπάθειας για ανθεκτικότητα υπάρχει ένα ε, αναβαθμισμένο σχέδιο, δράση, ε, σχέδιο δράσης για τον ε, χημικό, βιολογικό, ε, ραδιολογικό κίνδυνο κτλ. Ε, ο κίνδυνος βεβαίως ε, για τις επιθέσεις θεωρείται χαμηλός ακόμα, αλλά δεδομένες της ε, του υλικού που, για το οποίο μιλάμε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι τρομοκράτες δεν έχουν πρόσβαση σε το υλικό ραδιολογικό, βιολογικό κτλ. Ε, με χάρη στι γνώσει, ε, στι δεξιότητε κτλ., η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει ένα πολύ πιο καλό πλαίσιο για να μειώσει τέτοιου τύπου απειλέ. Νομίζω ότι αυτέ οι δράσει ε, είναι χρήσιμε για, για τα κράτη-μέλη και υπάρχει και η χρηματοδότηση για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη προ αυτήν την κατεύθυνση. Πρόσφατε επιθέσει χρησιμοποίησαν ε, το TATP, ένα, ένα εκρηκτικό που είναι ένα όπλο που επιλέγει ο ISIS. Έχουμε ένα κανονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιορισμό της πρόσβασης ε, στους, ε, στις πρόδρομες ουσίες ε, που τις ανακατεύουν με εκρηκτικά για να φτιάξουν το τελικό εκρηκτικό μηχανισμό και είπαμε χθες ότι θα, πρέπει να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια για να ενισχύσουμε την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού, τόσο ώστε να εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη, ε, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται και ταυτόχρονα να ξεκινήσουμε μία απλή αναθεώρηση του κανονισμού αυτού καθεαυτού με τα κρατημέλη για να ελέγξουμε κατά πόσον είναι κατάλληλος δεδομένου του επίπεδου απειλή. Ε, οι τρομοκράτε επίση δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα στατικά που χρησιμοποιούν για να φτιάξουν εκρηκτικά ε, και παράλληλα θα πρέπει να του αφαιρέσουμε και άλλα μέσα που χρησιμοποιούν στι επιθέσει. Χρησιμοποιούν ακόμα ε, τα μέσα επικοινωνίας, ε, ε, κρυπτογραφημένα μέσα επικοινωνίας επίσης, μεταξύ άλλων. Ένα πρακτικό βήμα που προτείναμε δεν είναι για να λύσουμε το θέμα της κρυπτογράφησης, το ευρύτερο θέμα. Ξέρετε ότι η κρυπτογράφηση είναι βασική για την ασφάλειά μας. Είναι κεντρικό στοιχείο του πακέτου που προτείναμε πρόσφατα για την ασφάλεια. Η θέση της Κομισιόν είναι ξεκάθαρη. Δεν μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε συστημική συστημικά, τις συστημικές, ε, συστημικά αναχώματα, αλλά μπορούμε ε, να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, του να χρησιμοποιείται η κρυπτογράφηση ως όπλο των τρομοκρατών. Εάν υπάρχει ένα υπολογιστής, ας πούμε, ή ένα τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, κάποια κράτη-μέλη είναι πιο ικανά να βρουν πληροφορίες από ένα τηλέφωνο πούμε, που έχουν κατασχέσει. Ε, θέλουμε λοιπόν να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, ε, την τεχνική πραγματογνωμοσύνη που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών και θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε, να επανενισχύσουμε την γνώση και το δυναμικό σε επίπεδο Europol που είναι η βασική υπηρεσία που υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στο επίπεδο αυτό. Ε, ένα άλλο τομέα του πακέτου αφορά τη χρηματοδότηση της δημοκρατίας ε, το σχέδιο δράση του 2016 για τη χρηματοδότηση της δημοκρατίας ε, είναι σχεδόν 100% σε εφαρμογή. Πρέπει να γίνουν ακόμα κάποια μικρά βηματάκια. Ένα όμως, ε, ένα βήμα για περαιτέρω δράση είναι η διασυνοριακή πρόσβαση τη χρηματοδότηση. Είναι, είναι βασικό θέμα στις έρευνες. Προσπαθούμε να δούμε ποια νέα μέρα θα μπορούσαμε να περάσουμε, τόσο ώστε οι αρχές να εντοπίζουν εάν ουσιαστικές, ε, στοιχεία για ουσιαστική χρηματοδότηση ε, τρομοκρατών ε, υπάρχουν σε άλλο κράτος μέλος. Οι πρόσφατες επιθέσεις από μοναχικούς λύκους μας υπενθύμησαν, λες και το θέλαμε, τη σημασία του να αντιμετωπίσουμε το βασικό πρόβλημα τη ρίζα του προβλήματο, τη ριζοσπαστικοποίηση. Έχουμε ε, μια ομάδα υψηλού επίπεδου ε, στην Κομισιόν για τη ριζοσπαστικοποίηση, με εκπροσώπου τη Επιτροπή σα επίση. Ε, και ελπίζω η ομάδα αυτή να κάνει συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς θα αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ρίζα του κακού, τη ριζοσπαστικοποίηση μέχρι το τέλος του 2017. Το ίντερνετ ήταν και παραμένει το βασικό εργαλείο για το ISIS για να ε, ξαπλώσουν την ε, νοσηρή τους προπαγάνδα και χρησιμοποιούν και αυτή την πλατφόρμα για να στρατολογήσουν κόσμο και να ε, κινητοποιήσουν τον κόσμο δράση ως μοναχικός λύκος. το G20, το G7, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν προωθήσει δράσεις σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε ό,τι μπορούμε όλο και περισσότερο στα πλαίσια του Φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εν ώψη του, της συνάντησης του Δεκεμβρίου για να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο με τους μεγάλους φορείς του ίντερνετ ε, αλλά και με μικρότερες πλατφόρμες, γιατί δεν μπορείς να λειτουργείς μόνο με τις μεγάλες. Εάν, ας πούμε, κατέβουν αυτές οι πλατφόρμες, ε, η κίνηση γίνεται αλλού. Έχουμε 50 διαφορετικές πλατφόρμες και κινούμαστε σε όλα τα επίπεδα και δραστηριοποιούμαστε σε όλα επίπεδα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να σημειώνουμε γρήγορη πρόοδο, καθώς και για τα αυτοματοποιημένα μέσα ε, εντοπισμού και κλεισίματος πολύ γρήγορα, αν όχι πρόληψη, α πούμε, του φορτώματο τέτοιου υλικού, με βάση τι πολύ σημαντικέ συζητήσει που είχαμε μέχρι στιγμή. Όπω ξέρετε όμω, μετά το, την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, έχουμε το δικαίωμα να αξιολογήσουμε την πρόοδο ε, αρχέ του 2018 και αν η πρόταση είναι αρκετά να δούμε τη δυνατότητα τότε για πιθανή νομοθεσία. Επίσης, ε, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τι οργανώσει κοινωνία των πολιτών, καθώ και άλλε φωνέ, οι οποίε ε, ε, μιλάνε με ένα τελείω διαφορετικό αφήγημα, αντίθετο από το αφήγημα τη Ομοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό για να κερδίσουμε τα μυαλά και τι καρδιές των ανθρώπων και να τους αποτρέψουμε από τη βία, από τον δρόμο της βίας, από την ατραπό της βίας. Στι αρχές του Οκτωβρίου ε, ξεκίνησαμε μια πρόσκληση υποβολής διαγωνισμού για την ενίσχυση της ε, κοινωνίας των πολιτών για να υπάρξει ένα αντιολικό. Το τελευταίο ε, πόδι του, ο τελευταίος πυλώνας είναι η συνεργασία. Ε, Εκ των όνων κάνε δεδομένε παγκόσμια απειλή που αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπέγραψε την ε, σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη τον Οκτώβριο του 2015 για την πρόληψη τη τρομοκρατία. Ε, θα πρέπει να τα επικυρώσουμε. 23 κρατημέλη όμω το έχουν κάνει. Το επιπλέον πρόσθετο στη σύμβαση έχει διατάξει για να γίνει πιο εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών και υπάρχει και κοινή απόκριση για να καταπολεμήσουμε του ξένου μαχητέ. Η επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμβαση και του Πρωτοκόλου θα είναι βασικό στοιχείο για να υποστηρίξουμε την, ε, τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ε, τώρα οι συνομοθέτες ε, μπορούν να προχωρήσουν με την ε, επικύρωση. Για να ενισχύσουμε τη συνεργασία της Europol με τρίτες χώρες, συστήνουμε στο Συμβούλιο να ανοίξει τις επραγματεύσεις ε, για ενίσχυση, ενισχυμένη συνεργασία με την Αλγερία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορτανία, Λίβανο, Μαρόκο, την Ισία και Τουρκία. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για το πόσο εύκολα θα είναι οι διαπραγματεύσεις αυτές ορισμένε μπορεί να είναι και περίπλοκε, γιατί όλοι ξέρουμε τα πρότυπα τα οποία θα εφαρμόσουμε, αλλά ξέρω ότι είναι σωστό να προσπαθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τη φύση της συνεργασίας μας με τις χώρες αυτές ε, της γειτονίας μας, που αντιμετωπίζουν επίσης ε, ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας, ε, γιατί καθώς το ISIS και το Χαλιφάτο περιορίζεται στο Ιράκ και στη Συρία. Χθες η Κομισιόν υπέβαλε συστάσει προ το Συμβούλιο για να ξεκινήσει την έναξη διαπραγματεύσεων για αναθεωρημένο PNR με τον Καναδά, ε, που το παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυ εσεί στην Επιτροπή σα. Όπω ξέρετε, ε, η απόφαση του δικαστηρίου τέλο Ιουλίου είπε ότι η προτινόμενη πρόταση PNR δεν μπορεί να ολοκληρωθεί υπό την τρέχουσα μορφή γιατί διάφορε διατάξει θεωρούνται ασύμβατε με τα πρότυπά μας, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και όπως είπα και στο παρελθόν, πρέπει να διατηρήσουμε ψηλά αυτά τα πρότυπα, αναγνωρίζοντα παράλληλα ότι τα δεδομένα PNR είναι βασικό εργαλείο στην καταπολέμηση τη δημοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματο. Επομένω, ε, υπάρχει αυτή η εντολή ε, και όταν εγκριθεί από το Συμβούλιο θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει με τον Καναδά, το στομότερο δυνατόν, για να θεωρήσουμε την ισχύουσα συμφωνία και να την ευθυγραμμίσουμε με όλε τι απαιτήσει που προβλέπει το δικαστήριο χωρίς να επηρεάσουμε άλλα στοιχεία της συμφωνίας. Αυτή η Επιτροπή παρακολουθεί το θέμα εδώ και καιρό και έχετε στείλει ένα ερωτηματολόγιο για το θέμα αυτό προς την Κομισιόν, το οποίο, στο οποίο έχουμε απαντήσει για πρώτη φορά χθε, πρώτη δέσμη απαντήσεων, με βάση τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση που κάνουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό μαζί σας. Η πρόοδος έχει κινήσει την καταπολέμηση του ISIS επιτόπου στο Ιράκ και στη Συρία ε, και αυτό είναι πολύ θετικό νέο. Καθώς χάνουν όμως έδαφος στις, στο λεγόμενο χαλιφάτο, δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι η τρομοκρατική απειλή θα μηδενιστεί. Το ISIS κοιτάει όλο και περισσότερο άλλους τρόπους για να λειτουργήσει, για να εξαπλώσει την προπαγάνδα του και να κάνει αυτό τον πόλεμο εναντίον στις αξίες μας και τον τρόπο ζωή μα. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση. Το πακέτο των προτάσεων που υιοθετήσαμε χθε είναι ένα τμήμα της απάντησης αυτό. Δεν πρόκειται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά ελπίζω ότι θα κάνει μια θετική συνεισφορά για να στα κράτη-μέλη ε, και στις αρχές των κρατών μελών που είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε King. Ε, ο Κλοντ Μωρά έπρεπε να φύγει για τη διάσκεψη των Προέδρων ε, σε σχέση με το Δουβλίνο και την ψηφοφορία που μόλις είχαμε. Οπότε ε, μην το πάρετε στραβά. Θα προεδρεύσω εγώ. Να περάσουμε σε, μια σε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές. Πρώτα το ΕΛΚ. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρομπέρτα και εκείνη έπρεπε να φύγει. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το, την ενημέρωση και την ανακοίνωση ε, για την τρομοκρατία. Χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερος και περιμένουμε εναγωνίως την εφαρμογή. Όσον αφορά τώρα το PNR Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, έχω μερικές ερωτήσεις θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι περισσότερο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, αν το έχετε υπόψη σας, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, πόσος χρόνος ε, θα χρειαστεί ακόμη για τις νέες διαπραγματεύσεις με τον Καναδά και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου βρισκόμαστε στο μεταξύ. γιατί η παλιά συμφωνία δηλαδή εξακολουθεί να ισχύει για όσους ταξιδεύουν στον Καναδά και πόσο είναι αυτό μια λύση ε, που να ε, μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Καταλαβαίνω ότι μιλώ με Βρετανό, αλλά τι, ε, τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, αν ο Καναδάς κάποια στιγμή πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε. Έχουμε τις δικές μας προδιαγραφές, θέλουμε να παραμείνουμε στις δικές μας προδιαγραφές. Υποχωρήσαμε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα άλλο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, ποιο είναι το σχέδιο, το εφεδρικό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και πάλι τον Επίτροπο ε, Κίνγκ. Ε, λέει η κυρία Σίπελ, ε, έρχεστε ε, συχνά στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να επιμείνω λιγάκι στην απόφαση του δικαστηρίου και την συνέχιση αυτή σε σχέση με το PNR. Τι θα γίνει αν ο Καναδάς επιμείνει ότι έχει τις δικές του προδιαγραφές και ότι δεν θέλουμε να τις αλλάξουμε. Και εμείς θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο, ότι επιμένουμε και εμείς ε, στις δικές μας προδιαγραφές. Ε, δεν ε, ε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πάντοτε να παρεκκλίνει από τις δικές της προδιαγραφές. Θα πρέπει να υπάρχουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αναφερθήκατε επίσης σε κάποιες πρώτες απαντήσεις από πλευράς Επιτροπής για τις δικές μας ερωτήσεις. Να σας πω την αλήθεια όμως, οι απαντήσεις αυτές είναι κάπως αόριστες για να το πω έτσι. Όταν πρόκειται λοιπόν για τη συμφωνία PNR με την Αυστραλία, ξέρουμε ότι ε, είναι επταετής και αν θέλουμε να την σταματήσουμε πρέπει να το κάνουμε το 2018, αλλιώς από το 2019 θα συνεχίσει για 7 ακόμη έτη. Αν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι πρέπει να το πούμε τώρα και πρέπει να κάνουμε νέα διαπραγμάτευση τώρα. Γιατί αν αναλύσουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξει, χάνουμε την ουσία και ενδεχομένως ε, μια λανθασμένη συμφωνία θα συνεχίσει να ισχύει. Ποιο είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμά σα ε, για να δούμε κατά πόσο χρειάζεται να αλλάξει κάτι και σε ποια χρονική στιγμή. Γιατί αν θέλουμε να την τροποποιήσουμε από κοινού με την Αυστραλία, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε σύντομα. Ένα ακόμη ερώτημα αφορά το PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέτε εσείς ότι τα κράτη-μέλη έχουν υποχρεώσει προκύπτουν από τις οδηγίες και λέτε ότι παραμένουν αναλύωτε. Αν προ, ε, συγκρίνω το κείμενο το PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με ε, του Καναδά σε σχέση με την περίοδο διατήρησης, για παράδειγμα. Εγώ βλέπω την ανάγκη αλλαγής του κειμένου. Τι ακριβώς λοιπόν θα σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Και τελευταίο σημείο, ενδεχόμενες συνέπειες σε, για άλλες αποφάσεις, όπως για, το, για παράδειγμα το σύστημα εισόδου-εξόδου στην απάντησή σας, λέτε ότι η νομική υπηρεσία έχει επιβεβαιώσει ότι αυτή η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν έχει αυτόματη, άμεση αυτόματη συνέπεια. Ε, δηλαδή υπάρχει έμεση. Τι εννοείται ακριβώς. Ε, ποιο είναι το αποτέλεσμα, γιατί σε σχέση με το F νομοθετήν ε, θα έπρεπε να ε, γίνεται μία ανάλυση όταν παραμένουν εκκρεμή ερωτήματα και ανησυχίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κανένας από το ECR που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Όχι, ωραία. Τότε φιλελεύθερη, κυρία Γκρίνσπεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με αυτό που είπατε, με αυτό που είπατε ε, προηγουμένως, ε, το, το σύνολο ε, των απαντήσεων σε σχέση με το κείμενο που ενέκρινε χθε το Σώμα των Επιτρόπων, θα έπρεπε να μην μας διαφεύγει ότι οι πολίτες μας θέλουν περισσότερο να γίνονται σε σχέση με την ασφάλεια ε, εντός της Ένωσης. Είπατε κάτι εχθές, το Ευρωβαρόμετρο είπε ότι ε, από το Ευρωβαρόμετρο προκύπτει ότι για τους πολίτες αυτό είναι το νούμερο ένα ανησυχία, η τρομοκρατία. Αυτή η τάση λοιπόν, σε σχέση με αυτό που είπατε εσείς για την τρομοκρατία, επιβεβαιώνεται και ε, σε επίπεδο Ευρωπαίων πολιτών, μια και το δείχνει το Ευρωβαρόμετρο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η παρουσίαση που μας κάνετε, γιατί αυτή η τρομοκρατική απειλή εξελίσσεται, είναι μόνιμη, είναι διασυνοριακή ε, και οι πολιτικές δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν σύνορα, πρέπει και αυτές να είναι ε, διασυνοριακές. Δεν πρέπει δηλαδή να σκεφτόμαστε σε ε, επίπεδο ε, κράτους μέλους μόνο, γιατί έχουμε μια κοινή ευθύνη. Δεν μπόρεσα να λάβω γνώση της των 80 σελίδων που περιλαμβάνει το πακέτο. Έχω όμως δύο-τρεις ερωτήσεις πολύ σύντομες. Πρώτον, επικροτώ τα 18,5 εκατομμύρια για την προστασία των δημοσίων χώρων ε, και την υποστήριξη των κρατών μελών και ε, των πόλεων. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, είναι πόλεις, είναι ε, χώρες που θέλουν να το κάνουν αυτό. Όχι ως χώρα η Γαλλία, οι πόλεις όσον αφορά αθλητικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. Και επικροτώ επίσης την ευαισθητοποίηση όλων των φορέων για την εξασφάλιση αυτής της προστασίας. Θα ήθελα όμως, και αυτό είναι μια, προ... μια πρόταση δύσκολη, αλλά δεν είναι παγίδα. Μας ρωτάτε πώς έχετε, πώς έχετε σκοπό ε, οι πολίτες να αποτελέσουν φορείς ε, ε, συμμέτοχοι της ίδιας τους της ασφάλειας. να μην είναι σε ένα σύστημα καταγγελία συνεχώς του τι συμβαίνει, κάτι που συμβαίνει τελευταίως λίγο χώρα, στη χώρα μου, σε μια περίεργη περίοδο. Λοιπόν, ε, αυτή η ιδέα λοιπόν της συλλογικής ε, ευθύνης ε, και της συλλογικής ασφάλειας, πώς έχετε σκοπό να την εφαρμόσετε ώστε να αισθάνεται μεμονωμένα ο κάθε πολίτης πιο ασφαλής. Κάτι ακόμη, η 11 έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια λέτε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Συμφωνώ να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση της ε, πληροφόρησης, ε, το είπε αυτό ο ίδιος ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, συμφώνησαν κάποιοι αρχηγοί κρατών ε, και κυβερνήσεων, όμως φοβίζει πάρα πολλούς άλλους ε, ηθήνοντες. Πώς λοιπόν έχετε σκοπό να γίνει η εφαρμογή αυτής της οντότητας, όπως και αν την αποκαλέσουμε, σε σχέση με μια φιλοσοφία κοινοτική προστασία των πολιτών κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και κάτι ακόμη. Μόλις ε, δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ενισχυμένη συνεργασία, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να παραταθεί η αρμοδιότητά του για την ε, εγκληματικότητα μεγάλης κλίμακας σε διακρατικό επίπεδο και να λαμβάνεται υπόψη μεταξύ αυτής και η τρομοκρατία. Δεν υπάρχει κανείς από την ΚΟΕ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Σαρτζεντίνη από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το PNR, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και PNR, αλλά και γενικώ για τα PNR. Τα αφήνω σε εσά, κύριε Πρόεδρε, είστε πολύ καλύτερο σε αυτά. Επίτροπε King, εκθέσει προχθέ ε, που έπεσε η Ράκα. Οπότε ε, βλέπουμε ότι το ISIS ε, όλο και περισσότερο παραγωνίζεται ε, και απομακρύνεται όλο και περισσότεροι ξένοι μαχητές, ντόπιοι, προσπαθούν να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και παιδιά που γεννιούνται στην περιοχή αυτή. Βλέπουμε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γίνονται από τζιχαντιστές που γυρνούν από τις περιοχές αυτές. Ε, εσείς ε, τι έχετε σκοπό. Υπάρχει μια πολιτική που να προβλέπετε για τα 28 κράτη-μέλη ε, και ποια ε, μορφή συνεργασίας ε, μπορούμε να σκεφτούμε. Γιατί στη δική μου χώρα, για παράδειγμα, αν υπάρχει διπλή υπηκότητα, να τους πάρουμε τη μία, κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν είναι υγιής τρόπος να αντιμετωπίσουμε, γιατί έτσι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι ξεκρέμαστοι σε άλλα σημεία του κόσμου που μπορούν μπορεί να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Άλλοι θέλουν τζιχαντιστές να τους ε, δικάσουν και να τους βάλουν ε, στα, στις φυλακή. Άλλοι θέλουν να τους επανεντάξουν. Είναι πολύ διαφορετικές οι προσεγγίσεις των κρατών μελών ε, για την αντιμετώπιση όσων επιστρέφουν από το ISIS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πολιτικές λοιπόν προβλέπουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές και με το γεγονός ότι πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, Κριστίνα Βίμπεργκ, για το EFTD. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επίτροπε, για την παρουσίασή σας. Σήμερα θα μιλήσω σουηδικά. Σε σχέση με το PNR, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος ε, ανταλλαγής πληροφοριών αν υπάρχει κάποια ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των ε, ε, ε, ταξιδιωτών, όσων ταξιδεύουν με αεροπλάνο, Είπατε επίση ότι θα υπάρξουν 100 εκατομμύρια από τα περιφερειακά ταμεία για την προστασία των δημοσίων χώρων. Πολύ καλά είναι όλα αυτά. Αλλά για ποιο λόγο είναι αυτές οι περιφέρειες τόσο ανασφαλής στην ε, Σουηδία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν στη χώρα μας, δεν παίρνουν άσυλο, δεν παίρνουν υπηκότητα και έχουν έναν αρκετά καταστροφικό τρόπο ύπαρξης, για να το πω έτσι, και ε, πρέπει να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν ε, και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η ριζοσπαστικοποίηση των ανθρώπων αυτών. Και να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα αίτια Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι στη Σουηδία οι οποίοι ε, βρίσκονται στο νοσοκομείο γιατί έχουν υποστεί τραύμα από, ε, από συγκρούσεις ε, ένοπλες. Πολλοί είναι όντως άνθρωποι που επιστρέφουν από χώρες όπου δραστηριοποιείται το ISIS και δεν υπάρχει επαρκής κατάρτιση στη Σουηδία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες χώρες κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις ε, και έχουν διπλή υπηκότητα θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η ευρωπαϊκή τους υπηκότητα και να ε, απομακρυνθούν γιατί πρέπει καταρχήν τους ε, πολίτες της χώρας μας ε, πρώτα να προστατεύουμε και νομίζω ότι αυτό μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών θα μας βοηθήσει σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ΕΝΕΦ δεν είναι παρούσα οπότε πηγαίνουμε στα υπόλοιπα μέλη των επιτροπών. Ινετφέλτ, Τζίνετζι, Βοσμάιερ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, κυρία Ινετφέλτ. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Έχω μια σύντομη ερώτηση για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για το PNR Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Ε, αναφερθήκατε σε μεγάλο βαθμό σε ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία μεγαλύτερη κλπ. Συμφωνώ, αλλά τι γίνεται αν ένα κράτο μέλο ή και περισσότερα κράτη-μέλη θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει ανεξάρτητη δικαστική εξουσία, όπω συμβαίνει στην Πολωνία για παράδειγμα. Πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών θα ανασταλεί με τη συγκεκριμένη χώρα ή θα λειτουργήσουμε, θα συνεργαστούμε με μία μη ανεξάρτητη δικαστική εξουσία. Για το PNR Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά λάβαμε μία απάντηση με την υπογραφή του κυρίου Τίμερμαν σήμερα και μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί είναι μια πολύ ατελής απάντηση, καθόλου πλήρης. Ε, μιλήσατε για την συνεχή ανάλυση της κατάστασης. Ε, η γνωμοδότηση όμως ε, εκδόθηκε στις 27 Ιουλίου. Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τότε και Εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι κανεί πυρηνικό φυσικό για να καταλάβει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι με ε, το PNR με τον Καναδά, αλλά και με τι Ηνωμένε Πολιτείε και με την Αυστραλία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν μια ολόκληρη στρατιά νομικών και πολύ ε, λαμπρών ανθρώπων που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα. Ο κύριος Τίμερμανς συμπεραίνει ε, ότι η νομική βάση είναι καλή για την ε, μεταφορά πληροφοριών στον Καναδά ε, κάποιος όμως πιστεύω ότι θα τον φυσβετήσει αυτό ε, στο δικαστήριο και μπορώ ένα πολύ καλό μπουκάλι σαμπάνιας ε, να το στοιχηματίσω λέγοντας ότι θα το χάσει, θα τη χάσει τη δίκη αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση PNR δεν υπάρχει νομική βάση, δεν υπάρχει συμφωνία και ακόμη και οι Ε, ε, συμφωνίες ε, ή εν πάση περιπτώσει ε, όταν στο λόγο μας ε, βασιζόμαστε για τέτοιου είδους ανταλλαγή απόψεων, δεν αρκεί αυτό. Η οδηγία αυτή τη στιγμή για το ευρωπαϊκό PNR ε, ικανοποιεί όλα τα κλητήρια που θέτει το δικαστήριο. Ο κύριος Τίμερμανς λέει, δεν απαντάει, λέει απλώς ότι συνεχίζει να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή της οδηγίας ε, για το PNR της Ένωσης. Ε, δεν λέει τίποτα αυτή η απάντηση, δεν λέει καθόλου κατά πόσο η οδηγία πληρεί τα κριτήρια ή όχι. Δεν υπάρχει απάντηση ουσιαστικά όσον αφορά τον αντίκτυπο στις συμφωνίες με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Αυστραλία. Αν το 2018 κατά τύχη έχουμε μία αυτόματη αναθεώρηση της επταετούς συμφωνίας, πολύ καλά. Αλλά αν δεν γίνει η αυτόματη αναθεώρηση, θα έπρεπε να τροποποιήσουμε τις συμφωνίες αυτές, γιατί είναι ηλίου φαϊνότερον ότι... Ε, η... Εντάξει, με την Αυστραλία μπορεί να διαφορετικά τα πράγματα, αλλά με τι ΗΠΑ όντω δεν πλήρει τα κριτήρια η συμφωνία. Και τέλος, ε, σε σχέση με το ευρωπαϊκό PNR, έχω ζητήσει πρόσβαση στα έγγραφα ε, σε σχέση με τα στοιχεία επαφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάθε εταιρεία που ενδιαφέρεται ή συμμετέχει στην εφαρμογή του ε, PNR της Ένωσης. Έχουμε πάρα πολλά χαρτιά στη διάθεσή μας και υπάρχει ένα, μια συγκεκριμένη ανταλλαγή email με μια συγκεκριμένη εταιρεία, την IBM, που δείχνει ότι αυτή η εταιρεία έχει σαφές συμφέρον όσον αφορά ε, την ε, έγκριση της συμφωνίας PNR και είναι σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι περιμένει την έγκριση για να αρχίσει να να ισχύει η συμφωνία. Ε, κάποια email δεν έχουν αποκαλυφθεί όμως. Ε, βέβαια ο διαμεσολαβητής το ελέγχει αυτό. Θα ήθελα πάντως να σας ρωτήσω, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε, πέρα από τη νομική διαδικασία, ότι θα μας αποκαλύψετε τις πληροφορίες αυτές για να ξέρουμε τι ακριβώς πλαίσιο υπήρχε και επιπίας βάσεως σε σχέση με την ε, έγκριση της οδηγίας. Ευχαριστώ. <coughs> Uh, Ευχαριστώ πολύ τρία ακόμα μέλη και μετά θα δώσουμε το λόγο ε, στους εκπροσώπους της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου και μετά ο λόγος και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Τσινίτση έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κιν που ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας. Προσωπικά με, ε, με ικανοποιεί που σας ξαναβλέπω, γιατί το γεγονός ότι είσαστε εδώ δείχνει την προσοχή σας και τη δέσμευσή σας για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσετε και το πακέτο των προτάσεων για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία ε, που υπάρχει στην έκθεση για την ε, κατάσταση της ασφάλειας στην Ένωση. Η προλαλή μου μίλησε για, σας μίλησε για την ανάγκη των μέτρων για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Εγώ θα σταματήσω και θα σταθώ μόνο σε δύο-τρία σημεία ξεκινώντας από τις πρώτες ε, επιθέσεις στο Παρίσι, στον Πατακλάν, μέχρι τις πιο πρόσφατος. Ε, είδαμε ότι τροποποιούν οι τρομοκράτες το modus operandi. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να υιοθετήσουμε μια πολιτική πρόληψης. Και έχω στο μυαλό μου αυτό που είπατε κι εσείς για, την, ε, για το θέμα της μεταφοράς πόρων για παράνομους σκοπούς, ε, για τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας που γίνεται και μέσω του ίντερνετ. Παράλληλα, μιλάμε για υπάρχουν μηνύματα μίσους και τα λοιπά ε, και ιδέες μίσους που εξαπλώνονται μέσα από το ίντερνετ. Το θέμα είναι πώς θα παρέμβουμε στο μέλλον. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να φανταστούμε τι θα κάνουμε με θέματα κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, γιατί εκεί θα παίξει το χαρτί της ε, πρόληψης στο μέλλον και εκεί θα δώσουμε έμφαση στις μελλοντικέ ε, έρευνες. Ξέρουμε ότι οι διοκτικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές έχουν δυσκολία να εντοπίσουν ε, κρυπτογραφημένες πληροφορίες ή να τις ε, διαβάσουν. Ειδικά όταν πρόκειται για Πληροφορίε που, έρχονται, που είναι σε τρίτες χώρες. Ε, θα χρησιμοποιούν και περισσότερο αυτό το μέσο οι τρομοκράτε. Τι νομοθετικά μέτρα μπορεί να προτείνει η Κομισιόν, ούτω ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση, τη διασυνοριακή πρόσβαση των αρχών σε τέτοιες ηλεκτρονικέ πληροφορίες. Η Κομισιόν πώς θα προωθήσει το διάλογο μεταξύ των δημοσίων αρχών και των, και των ιδιωτικών φορέων, ούτω ώστε ακριβώ να διευκολύνει τέτοιου τύπου έρευνε. Για το θέμα τη κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση πάλι, εγώ επισκέφθηκα την Europol πριν λίγε μέρε. Και διαπίστωσα ότι η Europol είναι ένα πολύ προηγμένο κέντρο ε, που ασχολείται με την αποκρυπτογράφηση. Εσείς ε, υπενηχθήκατε σε αυτό το αυτό το πράγμα μέσω των καλών πρακτικών, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Κομισιόν τη Europol, γιατί ξέρετε ότι ειδικά για την αποκρυπτογράφηση χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις ε, για να έχουμε την κατάλληλη πληροφορική. Και δεν μπορούν όλες οι χώρες να, πάρουν, να αγοράσουν αυτό τον εξοπλισμό, αυτές τις τεχνολογικές δομές. Πώς λοιπόν σκοπεύει να βοηθήσει η Κομισιόν. Τελευταίο σημείο που νομίζω ότι είναι τεράστια σημασία και για σας, το θέμα της ρεσπαστικοποίησης, το αναφέρατε κι εσείς. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία. Τι μπορεί να κάνει τώρα η στιγμή σε ό,τι αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση και κυρίως τη ριζοσπαστικοποίηση ε, στο χώρο των φυλακών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σον Μάιερ τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Χολμάιερ, μετά τα όσα ανέφερε η κυρία Κινίτσι, βλέπουμε ότι σε ό,τι φορά το προσωπικό της Europol κάνουμε πολύ μικρά βήματα. Εντάξει, κάπως ε, σημειώνουμε πρόοδο, αλλά εάν λάβουμε υπόψη τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει ενώπιον των 28 κρατών μελών, καλό θα ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση και με πιο πλούσιο περιεχόμενο και όχι μόνο μία-δύο φορές το χρόνο. Θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες από ε, τη Διευθύνουσα Επιτροπή πιο συστηματικά. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν και επαρκές προσωπικό για να καλύψουν όλες τις αρμοδιότητες. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την επαρκή στελέχωση του οργανισμού για να πεταχύνουμε έτσι τις διαδικασίες και να βεβαιωθούμε ότι ε, εκπληρώνονται όλες τις αρμοδιότητες γιατί έχουν και την καταπολέμηση της δημοκρατίας, τις ε, ενέργειες κατά της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Και συνεχώς έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλη έλλειψη προσωπικού και νομίζω ότι αυτό δεν επιτρέπει στον οργανισμό ε, να παρέχει τη στήριξη που θέλει και πρέπει προς τα κρατη Αυτό είναι το πρώτο. δεύτερο. Η Τουρκία στέλνει αυτή τη στιγμή δεδομένα στην Interpol για μεμονωμένα άτομα με βάση το δικό τους ε, αρκετά ιδιαίτερο ορισμό της τρομοκρατίας. Και υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκράτες ε, στην Ισπανία και αλλού μόνο και μόνο επειδή διαφωνούν πολιτικά με τον κύριο Ερντογάν. Ανεξάρτητα αν αυτά τα άτομα μου αρεστά ή όχι, Θεωρώ ότι ο ορισμός της τρομοκρατίας θα πρέπει να θεσπιστεί από την Interpol. Να μην χαρακτηρίζει δηλαδή κάποιο απλό πολίτης μιας ξένης χώρας ω τρομοκράτης βάσει αυτού του ιδιαίτερου ορισμού και περίεργου ορισμού. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ενιαίο ορισμό της τρομοκρατίας στην Interpol ήταν καλό να υπάρχει αυτό. Και κάτι τελευταίο. Αναφέρατε ορισμένους πόρους που θα δώσατε για την προστασία των δημοσίων ε, χώρων. Ε, θα έπρεπε να υπάρχει μια εξολόγηση αντικτύπου ε, και μπορεί να υπάρχουν περιπτώσει όπου μιλά... κάνουν λόγο για έναν ενδεχόμενο κίνδυνο, αλλά όχι πολύ μεγάλο κίνδυνο. Οπότε ίσως σε κάποιες περιοχές χρειαζόμαστε πιο σύγχρονες μεθόδους για να αποτρέψουμε αυτές τις ενέργειες ε, και για να στηρίξουμε τις αστυνομικές αρχές. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σε αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Ζήπελ. Ξέχασα κάτι. Να πω κάτι όμως πρώτα για το προσωπικό της Europol. Συμφωνώ σε αυτό. Το πρόβλημα όμως ξεκινάει από τα κράτη-μέλη, θεωρώ. Γιατί και στις αστυνομικές μας αρχές ε, υπάρχει υποστελέχωση. Και κάποιες φορές δεν υπάρχει και επαρκής εξοπλισμός. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο ε, τα περισσότερα κονδύλια. Πρέπει σε ε, εθνικό επίπεδο να διαπιστεύσουμε περισσότερους αστυνομικού, ούτω ώστε αυτοί να συμμετέχουν και στι εθνικέ αστυνομικέ αρχέ και στη Europol. Για την κρυπτογράφηση. Εν τω μεταξύ όλοι λένε τι σημαντική που είναι η κρυπτογράφηση. Εντάξει. όμω εμένα με προβληματίζει λίγο αυτή η έκφραση ότι δεν θέλουμε να έχουμε ε, συστηματικά παραθυράκια. Δεν θέλουμε να έχουμε μη συστηματικά παραθυράκια. Δεν θέλω να επισέλθω τώρα στι τεχνικέ λεπτομέρειε. Κάποιο όμω ανέφερε ότι ίσως χρειαστεί συνεργασία με ιδιωτικέ επιχειρήσεις, ώστε να βρούμε ε, σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις βέβαια να βρούμε τρόπο αποκρυπτογράφησης αυτών των δεδομένων. Όμως, αν χρειαζόμαστε τη στήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων ή ε, μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το παραθυράκι, όποια μορφή και αν έχει, δεν θα αξιοποιηθεί ενδεχομένω μόνο από τι κυβερνητικέ αρχέ με ξεκάθαρα εχέγγυα και προποθέσει, αλλά αυτό το παραθυράκι θα υπάρχει και σε άλλου τομεί, ιδιωτικού. Οπότε η κρυπτογράφηση πια δεν θα έχει νόημα ακόμα και για τους καλούς και χρήσιμους ε, σκοπούς. Υπάρχει απάντηση. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στην Προεδρία του Συμβουλίου να σχολιάσει. Πριν από αυτό όμως, να επαναλάβω τα λόγια του συγκεκριτή για τις συμφωνίες PNR, για τις συνέπειες ε, της συμφωνίας ε, με τον Καναδά και στις άλλες ε, συμφωνίες για την οδηγία PNR. Υπάρχει αυτό το ερώτημα για την ε, διατήρηση των δεδομένων, αλλά και για το PNR. Αν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε πιο στοχευμένη διατήρηση, μέτρα στοχευμένη διατήρησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε εδώ και 10-15 χρόνια. Α, πρέπει να φύγω, λέει ο επίτροπο. Εντάξει, τότε να δώσουμε το λόγο πρώτα σε εσά. Και μετά στο, στην Προεδρία, αν δεν του πειράζει. Συγγνώμη. Αλλά για να μην έχω μόνο δύο λεπτά στο τέλος, Μπορεί να μην είμαι στη θέση να απαντήσω σε όλα σα τα ερωτήματα, αλλά θα προσπαθήσω, τουλάχιστον αφού έχω και λίγο περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ θετική όλη αυτή η έμφαση που δίνεται σε αυτό το ευρύ φάσμα ζητημάτων. Δεν νομίζω ότι θα μπορούμε να τα καλύψουμε όλα αυτά τώρα. Παραμένω βέβαια στη διάθεσή σα για να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσει. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη συνεργασία μα και εδώ και στην Ειδική Επιτροπή. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε πάντα 100%, θεωρώ ότι έχουμε επαγγελματικό διάλογο σε αυτά τα ζητήματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Υιοθετούμε μια σειρά μέτρων τα οποία έχετε θίξει για τους δημόσιους χώρους, τις εκρηκτικές ύλε, την κρυπτογράφηση, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που βασίζονται στη δουλειά που έχει ήδη γίνει. Εναρμόνιση των προτύπων σε όλα τα κράτη-μέλη, αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων για τα εξωτερικά σύνορα, την ανταλλαγή προφοριών, τις μυστικές υπηρεσίες ε, και τον κατάλληλο εξοπλισμό των οργανισμών μας, των υπηρεσιών μας για να στηρίξουν ε, ε, τα κράτη-μέλη. Κανένα από αυτά τα στοιχεία από μόνο του δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, την απειλή. Όμως από κοινού συμπληρωματικά αυτά τα μέτρα μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αυτό είναι το πνεύμα στο οποίο εμείς θέλουμε να κινηθούμε. Συμφωνώ με την κυρία Κιχρισμπέκ ότι ε, παραμένει υψηλή η ανησυχία ε, του, των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κάνουμε προσπάθειες ότι αφορά τον έλεγχο πληροφοριών στα εξωτερικά μας σύνορα ανταλλαγή πληροφοριών, στήριξη αυτής της ε, ανταλλαγής. Όλα αυτά έχουν να κάνουν εν μέρη και με την ε, απειλή που προκύπτει από τους Ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή τους που έχουν μεγαλώσει εδώ, όπως ανέφερε ο Πέρος Μακρόν χθες. Αλλά ο Ντάις βλέπουμε ο ότι παραμένει δραστήριος, ενεργός, ε, αποστέλλοντα μήνυμα από τη βάση στο Ιράκ και τη Συρία. Και χθε στο Σώμα των Επιτρόπων συζητήσαμε ακριβώ αυτή την ε, συνεχιζόμενη απειλή των αλλοδαπών μαχητών που επιστρέφουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Όμω αναγνωρίζουμε και την ε, απειλή ω προ την ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη, αλλά και ω προ ε, πολλέ από τι γειτονικέ μα χώρε εταίρου. Γιατί είπαμε ότι κάποιοι θα χαθούν, κάποιοι θα ε, πάνε αλλού για να συνεχίσουν την πάλη τους, όπως την αποκαλούν, και αυτό το αλλού μπορεί να είναι και οι γειτονικές μας χώρες. Πρέπει να δούμε εμεί πώ θα τηρήσουμε τα πρότυπα που έχουμε θέσει και να συνεχίσουμε τη συνεργασία και με τι γειτονικέ μα χώρε, τι χώρε εταίρου μα. Σε ό,τι φορά όμω την απειλή προ την ασφάλεια, αναμφίβολα ε, θέτει και ορισμένε κοινωνικέ ε, προκλήσει, όπω ανέφερε η κυρία Βίνμπεργκ είτε πρόκειται για τις ε, υπηρεσίες υγείας, είτε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια σε βάθος συζήτηση σε σχέση με τα όσα λέμε μέχρι σήμερα, γιατί θα κάνουμε με αυτούς που επιστρέφουν, που δεν ήταν όμως μαχητές. Για τους μαχητές υπάρχει συνένεση ότι θα ε, τους αναλάβει το δικαστικό σύστημα, η δικαιοσύνη. Όμως, γυναίκες, παιδιά, υπάρχει διαφορετική πρόκληση από ριζοσπαστικοποίησης και κοινωνικής επανένταξης και στηρίξή τους. Και για να είμαι δεν έχει ξεκινήσει σε βάθος ακόμα αυτή η συζήτηση. Καλά κάνετε λοιπόν και το φύγετε. αυτό το θέμα. Να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ρίζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο, όπως ανέφερε η κυρία Κινίτσι και είναι ένα από τα βασικά ε, θέματα της ε, διπλογικής διάσκεψης ε, G7 αύριο στην Ιταλία. Με αυτό έχει να κάνει και το θέμα της κρυπτογράφησης. Όπως αναφέρει η κυρία Σίπελ, η κρυπτογράφηση δεν αφορά μόνο την, μια καλή ισορροπία. Τι κάνουμε δηλαδή όταν έχουμε κατάσχεση μια συσκευή υπό πολύ συγκεκριμένε συνθήκες. Πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν περαιτέρω. Θέλουμε να βρούμε τρόπους πρακτικής στήριξης προς τις αρχές επιβολής του νόμου, ε, πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με συγκεκριμένε συσκευέ υπό πολύ αυστηρέ προποθέσει στο πλαίσιο ε, μια ε, ποινική έρευνα στο πλαίσιο καταπολέμηση δημοκρατία. Όμω πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και με την κρυπτογράφηση λοιπόν ευρύτερα στην επικράτειά μας αλλού. Θα το καλύψουμε αυτό το θέμα του χρόνου όταν λέμε ότι θα ενισχύσουμε τις προσπαθειές μας για τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Στήριξη προς τους οργανισμούς και υπηρεσίες μας ε, και στελέχωση που ανέφερε η κυρία Χολμάιερ, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Εγώ είμαι υπέρμαχος της Europol. Συνεχίζει να μεγαλώνει η Europol και με τη δική σας στήριξη. Έχουμε χρηματοδότηση για 86 επιπλέον θέσεις για του χρόνου. Εάν χρειάζεται παραπάνω πόρους η Europol, θα έρθουμε σε εσά και θα το συζητήσουμε. Δεν ε, θα είμαστε φιδωλοί με τη στήριξή μας προς αυτόν τον οργανισμό. Για το θέμα τώρα των μυστικών υπηρεσιών που ανέφερε η κυρία Γκρισμπέκ και άλλοι. Το σημείο εστίασή μα ε, σε αυτή τη δέσμη είναι τα επόμενα πρακτικά βήματα που θα κάνουμε. Γιατί όντω αυτή η συζήτηση πολύ γρήγορα παίρνει πολιτικές διαστάσεις και σε κάποιες φορές ε, οδηγεί και σε υπερβολική πόλωση. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πρακτικά ζητήματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι και έτσι να σημειώσουμε γρήγορα πρόοδο. Πρέπει να ενισχύσουμε τη χρήση του συστήματος ε, SIS, ανταλλαγή προφοριών Schengen. Ε, και να συμφωνήσουμε ότι όταν κάποιος συνδέεται με τρομοκρατία, να υπάρχει κοινοποίηση στο σύστημα SIS. Μου προκαλεί, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονό ότι δεν έχουν πρόσβαση όλε οι μυστικέ υπηρεσίε των κρατών μελών στο σύστημα SIS. Αυτό είναι παράξενο. Θα πρέπει λοιπόν να συνδεθούν όλες οι υπηρεσίες αυτές στο σύστημα SIS. Αυτά είναι πρακτικά. Πολύ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να κρύβουμε το γεγονό ότι υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ, συγγνώμη, και συνεργασία μεταξύ μυστικών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Υπάρχει. Πρέπει να δούμε πώ θα διαμορφώσουμε συνδέσμου και αλληλεπίδραση μεταξύ αυτή τη συνεργασία και των μυστικών μας υπηρεσιών, βασιζόμενοι και στην εθνική μας εμπειρία, αλλά βέβαια με σεβασμό προς τι εθνικέ ιδιαιτερότητε. Στηρίζω ε, την ε, άποψη που να δώσουμε περαιτέρω αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολύ χαίρομαι που έχουμε 20 κρατημέρια, πρέπει να συνεχίσουμε. Είχαμε λοιπόν μια σειρά θεμάτων που θίξατε που δεν είχαν σχέση με το PNR. Τώρα λοιπόν στρέφομαι στο PNR, γιατί δεν θα το αποφύγω. Α, όχι, δύο ακόμα. Πολωνία. Ξέρετε ότι έχει κοινωνική διαδικασία, γιατί είχατε και έναν ιδιαίτερα ζωντανό διάλογο με τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμαντς επί του θέματος. Νομίζω ότι ο Τίμερμαντς ελπίζει ότι θα σημειωθεί πρόοδος στο πλαίσιο διαλόγου που προτείνει. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να διατηρήσουμε την συνεργασία με τις πολωνικές αρχές για την αντιμετώπιση των απειλών. Ήμουν στη Βαρσοβία την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουμε την πρακτική συνεργασία που μπορούμε να έχουμε. Τουρκία και Ιντερπόλ. Δεν είναι μόνο θέμα της Τουρκίας Υπήρξαν και άλλα προβλήματα με τις κόκκινες ε, κοινοποιήσεις ε, μέσω της Interpol. Ξέρετε ότι με την αυστηρή έννοια του όρου δεν είμαστε μέλη της Interpol, όμως έχουμε ενεργό διάλογο για να ανοίξουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς ε, ανακύπτουν τέτοιες προκλήσεις που αναφέρατε. Τα διάφορα ερωτήματα που άκουσα για το PNR. Ε, ζητώ συγγνώμη που θεωρείτε ότι, είμαστε αργοί. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε να είμαστε διεξοδικοί απλώ. Έχουμε δώσει κάποιε πρώτε απαντήσει στα ερωτήματα μα που βάλατε γραπτό, γιατί θεωρώ ότι για λόγου σεβασμού θα πρέπει να έχετε γραπτέ απαντήσει στι γραπτέ σα ερωτήσει πριν με δείτε κιόλα με σάρκα και ωστά, Πριν μιλήσουμε διαζώσει αλλά αναγνωρίζω ότι οι γραπτές απαντήσεις δεν καλύπτουν όλα τα θέματα που θέσατε. Αξίζεται να σας δοθούν απαντήσεις, πλήρεις απαντήσεις και ελπίζω στη σημερινή συζήτηση και στις περαιτέρω επαφές μας θα δώσουμε τελικά απαντήσεις και θα αναγνωρίσουμε τις ορισμένες περιπτώσεις. Ίσως δεν θα μπορέσουμε ε, να... Μπορεί να μην σας πίσω 100% στις απαντήσεις μου, αλλά θα προσπαθήσω. Λοιπόν, Διαφορετικέ ερωτήσει ακούσαμε, θα προσπαθήσω να τις καλύψω όλες. Το χρονοδιάγραμμα του PNR. Έχουμε την εντολή, μάλλον την έχουμε υποβάλει, ελπίζω να εγκριθεί γρήγορα. Οι Καναδοί θα τους, θα τους δούμε στα πλαίσια του, του G7 σήμερα και αύριο και θα τους ενθαρρύνουμε και σήμερα και ξανά να πάρουν και την δική τους εντολή, ε, την επίσημη εντολή, για να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν τις συζητήσεις. Και θέλω να προχωρήσουν αυτές τις συζητήσεις γρήγορα. Παρότι θεωρώ ότι η βάση για τις μεταφορές δεδομένων είναι καλή. Μπορούμε να διαφωνήσουμε βεβαίως αυτό, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι. Συμφωνώ παρόλα αυτά ότι δεν θα πρέπει να κολλήσουμε. Θα πρέπει να υπάρξει νέα συμφωνία. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε τώρα να πετύχουμε νέα συμφωνία ε, που να ευθυγραμμίζεται με την γνωμοδότηση του δικαστηρίου. Κάτι άλλο τώρα. Εγώ δεν, θα πρέπει να δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάζουμε το σενάριο του να μην υπάρξει συμφωνία. Δεν συμφωνώ με αυτό. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία για την, τις άμεσες επιπτώσεις για άλλες διεθνείς συμφωνίες που θα έχει συμφωνία με τον Καναδά. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί η θέση μας με βάση την ανάλυση μας είναι ξεκάθαρη ότι άλλες συμφωνίες της Αυστραλίας, των Ηνωμένες Πολιτείες, οποιασδήποτε άλλες είπατε κι εσείς, ισχύουν μέχρι να ανασταλούν, τερματιστούν ε, αντικατασταθούν ή ακυρωθούν. Αυτή είναι η δική μας αξιολόγηση. Ξέρετε γιατί αναφερθήκατε σε αυτές ε, τους μηχανισμούς για την παράταση των συμφωνιών αυτών ή οποιαδήποτε άλλη τον τερματισμό τους ή οτιδήποτε. ξέρετε τι, ε, τι συμβαίνει το επόμενο καλοκαίρι και μετά θα πρέπει να συνεχίσουμε μετά το καλοκαίρι. Ε, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε κάποιες συμφωνίες. Υπάρχουν κάποια ορόσημα χρονικά, αλλά νομίζω θα πρέπει να τις επαναξετάζουμε. Επίσης αναγνωρίζω ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στις διάφορες συμφωνίες, γιατί υπόθηκε σε κάποιες ερωτήσεις, δεν είναι ακριβώς οι ίδιες, δεν είναι πανομοιότυπες. Για το θέμα της ε, αντιπαραβολής με τη Συμφωνία PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι είναι να λέτε ότι δεν έχουμε πάρει θέση σε αυτό. Ε, είπαμε και εγώ το είπα δημοσία και νομίζω ότι υπάρχει και γραπτό στο πακέτο μας ότι η άποψή μας είναι ότι οι υποχρεώσεις στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη που απορρέουν από την οδηγία PNR δεν επηρεάζονται από την γνωμοδότηση του δικαστηρίου. Μπορεί να διαφωνήσετε με αυτό, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστό να πείτε ότι δεν έχουμε πει θέση μα. Αυτή είναι η θέση που έχουμε καθορίσει και έχουμε εκφράσει. Πιστεύουμε ότι οι διαφορετικές νομικές καταστάσεις της ε, Οδηγίας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης PNR για τη συλλογή από τα κράτη-μέλη, την αποκλειστικά για τις διοκτικές αρχές και την εφαρμογή του νόμου και το γεγονός ότι δεν συνδέεται με διεθνείς συμφωνίες αλλά αφορά τις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και για την, τα ταξίδια στον χώρο Σέγγεν, τη θέτει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από τι υπόλοιπε συμφωνίε. Το συζητάμε βέβαια αυτό. Τώρα, για τα άλλα εργαλεία και το ερώτημα που ακούσαμε σχετικά με αυτό το θέμα. Είπαμε πολύ σύντομα, και κάποια στιγμή θα πρέπει να το πούμε και πιο μακροσκελώς, ε, ποια είναι η αρχική μας αξιολόγηση για την επίπτωση και τι επιπτώσει και τις ε, συνέπειε που θα έχει στα άλλα εργαλεία ε, που ζητάτε, που μας ρωτάτε. Λόγω της ε, διαφορετικής φύσης των εργαλείων, εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει άμεση επίπτωση. Δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο όμως σήμερα να συζητήσουμε διεξοδικά κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία, κάθε ένα από αυτά τα μέσα ε, και κείμενα, αλλά μπορούμε να την κάνουμε αυτή η συζήτηση. Πάντως, η υποκείμενη βάση της συζήτησής μας είναι ότι η απάντηση του δικαστηρίου στη γνωμοδότηση αφορά ένα συγκεκριμένο νομικό εργαλείο που αφορά μία συγκεκριμένη κατάσταση και τα απορίσματα της νομοδότησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτόματα σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό το επιχείρημα αφορά και άλλες αποφάσεις του δικαστηρίου σε άλλους τομείς. Ότι μιλάμε για συγκεκριμένες καταστάσεις και συγκεκριμένα νομικά πλαίσια. Κάθε μία από τις αποφάσεις θα πρέπει να ειδωθεί χώρια μέσα στο δικό της πλαίσιο σε χωριστή λεπτομερή συζήτηση μαζί σας. Κάνα πρόβλημα την κάνουν. Μέσα σε αυτό το πνεύμα λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας πάνω σε αυτό το φάκελο που, έχει, που πολύ προσοχή, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που, έχουμε, ε, μας έχουν απασχολήσει. Δυστυχώς πρέπει να φύγω. Δεν θέλω να αποφύγω τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε Κίν. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Επίσης, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Προεδρία του Συμβουλίου η Σόφιν Βέρτ επίσης θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Αλλά σύντομα παρακαλώ. Ή να το αφήσουμε, το ακούσουμε μετά την παρουσίαση του, της Προεδρίας του Συμβουλίου. Θέλεις τώρα, σύντομα Σόφι. Μου φαίνεται κοινικό. Δεν είναι παιχνιδάκι τώρα αυτό. Η στάση της Κομισιόν νομίζω ότι είναι περιφροντική και για το δικαστήριο και για τους πολίτες. Η Κομισιόν θα πρέπει να σεβαστεί τις συνθήκες. Δεν μπορείτε να βάλετε το άχθος στους επιμέρους πολίτες όπου κάθε φορά πρέπει να πηγαίνουν στο δικαστήριο και να ε, διεκδικούν πράγματα επί χρόνια. Ξέρετε πολύ καλά τι θα, κάνει, ε, θα συμβεί αν κάποιος αμφισβητήσει τη συμφωνία με τις ΟΠΑ στα δικαστήρια και προσφύγει στα δικαστήρια. Α μην παίζουμε παιχνιδάκι και προσποιούμαστε τώρα. Α, είναι διαφορετική συμφωνία, πρέπει να την κοιτάξουμε. Το ξέρετε πολύ καλά. Η Κομισιόν έχει την υποχρέωση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι αποδεκτό Ευρωπαίοι πολίτε να πρέπει να προσφύγουν στο δικαστήριο για να ασκήσουν τα δικαιώματά του, γιατί του εγκαταλείπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν μιλάμε για το διάλογο τώρα. Σίγουρα ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε για το θέμα του διαλόγου. Η Κομισιόν έχει ένα καθήκον να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και να διαφυλάξει τις συνθήκες. Και δεν το κάνει. Δεν κάνει το καθήκον της. Ναι, αναγνωρίζω ότι έχουμε αυτό το καθήκον. Και λογικό είναι να λέτε ότι πρέπει να κοδοτήσουμε σε σχέση με αυτό το καθήκον. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δείξω έλλειψη σεβασμού προ τη δική σας επιτροπή και τι υπόλοιπε επιτροπέ που ασχολούνται με αυτά τα θέματα αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το πνεύμα προσπαθώ να απαντήσω αυτά τα ερωτήματα. Σας ε, αφήνουμε εδώ να φύγετε. Ε, έχετε άλλες ε, ανηλυμένε υποχρεώσεις. Χαίρομαστε που έρχεστε συχνά να συζητάμε εδώ. Ο κύριος Τάιο, από την Προεδρία του Συμβουλίου, θα απαντήσει για τα ίδια θέματα. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, προσκαλείστε το Συμβούλιο σήμερα για να ανταλλάξουμε απόψει για την γνωμοδότηση του Συμβουλίου για την ενδεχόμενη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά για το PNR. Φυσικά είμαι ευγνώμων προς τον Επίτροπο Κίνγκ που απάντησε πολλές από τις ερωτήσεις σας και δεν ξέρω πόσο νόημα έχει να συμμετάσχει το Συμβούλιο, να πει το Συμβούλιο τη δική του άποψη για αυτό το θέμα τώρα. Ίσως το πιο σημαντικό που θα μπορούσα να σας πω και να δεσμευτώ σε σχέση με αυτό είναι ότι όπως σας εξήγησε και ο Επίτροπος Κίνγκ, η σύσταση προς το Συμβούλιο για να επαναδιαπραγματευτεί την εντολή μας παρουσιάστηκε χθες και ως εκπρόσωπος Προεδρίας επιβεβαιώνω ότι έχουμε την πρόθεση να εργαστούμε αμελητή. Οι ομάδες εργασίας θα ξεκινήσουν πάρα αυτά τη δουλειά και όπως ε, σας είπε και ο Επίτροπος Κιν, ελπίζουμε να υπάρξει μια γρήγορη εντολή. Από και πέρα είναι στο μπαλάκι της, ε, στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επαναδιαπραγματευτεί τη συνθήκη. Το Συμβούλιο έλαβε και ένα κατάλογο ερωτήσεων από το Κοινοβούλιο. Για λόγους συντομίας θα ασχοληθώ μόνο με τα πιο σημαντικά σημεία. Και ζητώ συγγνώμη αν θα υπάρξουν κάποιες επαναλήψεις. Μετά όσα είπε ο Επίτροπος. Uh, as concerning implications... Για τις επιπτώσεις της νομοδότησης του δικαστηρίου σε άλλες συμφωνίες. Η γνωμοδότηση ε, δεν αφορά συμφωνίες με άλλες χώρες. Είναι η νομική προσέγγιση. Θα πρέπει να την ε, ελέγξουμε. Αυτές οι συμφωνίες όμως εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που δεν έχουν ε, κηρυχθεί άκυρες από το δικαστήριο, δεν έχουν λήξει ή δεν τις έχουν επαναδιαπραγματευτεί τα μέρη των συμφωνιών αυτών. Το ίδιο ισχύει και για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το PNR. Είναι μια αρχή η οποία ισχύει και τη δέχεται και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, μέσω πολλών ε, υποθέσεων και αποφάσεων. Τα κράτη-μέλη νομικώ πώ είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία όπω έχει στην εθνική του νομοθεσία. Είναι ένα σαφέστατα δύσκολο καθήκον το οποίο προσπαθούν να εκπληρώσουν τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Τρίτον, πιθανές επιπτώσεις στην συνεχιζόμενη δουλειά που κάνουμε μαζί καθώς για αυτό το θέμα και για άλλους νομοθετικούς φακέλους. Αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική συμφωνία για το σύστημα εισόδου-εξόδου. Εμείς παρακολουθούμε την ε, γνωμοδότηση του... των νομικών υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων και συμφωνούμε. Είπαν ότι το κείμενο εισόδου-εξόδου ε, ικανοποιεί τις, ε, το τεστ αναγκαιότητας με βάση τα κριτήρια του δικαστηρίου. Η Ιστονική Προεδρία επικυρώνει πλήρως τη θέση των νομικών υπηρεσιών που θεωρούν ότι ο σκοπός του σχεδίου κανονισμού εισόδου-εξόδου είναι διαφορετικό από τη συμφωνία PNR με τον Καναδά. Και εδώ η φύλαξη των δεδομένων που προβλέπεται στο σχέδιο κανονισμού δεν αμφισβητεί σε καμία περίπτωση την νομιμότητα της πολιτικής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Μετά τα αυτά, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και θα να σας πω πρώτα ότι ε, με αυτά που είπα ούτως ή άλλως εξαρτήθηκε και ο χρόνος μου. I'm glad I'm... Παρακαλώ, καθίστε λιγάκι ακόμα. Ζητώ συγγνώμη που σας πιέζουμε χρονικά. Δεν βλέπω ερώτηση αυτή τη στιγμή. Ε, πάντως θα είμαστε σε επαφή για αυτό το θέμα. Ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε για τη σημαντική αυτή ανταλλαγή απόψεων. Και μετά τα αυτά συνεχίζουμε και πάμε στο επόμενο σημείο στη Μέση Διάταξη που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ε, λειτουργία και την διαχείριση μεγάλων συστημάτων πληροφορική στον τομέα της ελευθερία δικαιοσύνη και ασφάλειας. Η Μόνικα Μακοβέη. Θα ακούσουμε το, την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης για την αναθεώρηση του πλαισίου EU-LISA. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια καταρχήν και συνεχεία στους σκιώδεις ηγητές και στους βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Έχουμε μαζί μας και την, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, Πασκαλ Μίλο, ε, βοηθός του Ματάρχη από τη Γενική Διάθεση Home. Μπορεί να παρέμβει επίση. Πρώτα η κυρία Μακοβέη όμως. Thank you very much. So four years after uh, Ευχαριστώ. Χρόνια μετά το, την έναρξη ισχύω τη EU Λίσα πρέπει να ενισχυθεί στην, ε, στα καθήκοντά τη γιατί έχει να αντιμετωπίσει τι προκλήσει τη μετανάστευση αλλά και της τρομοκρατία. για την εξασφάλιση της ασφάλειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα με την πρόταση ευρωπαϊκή ε, Επιτροπής ε, ε, που διευρύνει κάπω το πεδίο αρμοδιοτήτων του eu θα έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη των συστημάτων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, του συστήματος εισόδου-εξόδου, του αιτία, του έκρης, δηλαδή για το ποινικό μητρό και το DCN, Όπω επίση ε, ο συγκεκριμένο οργανισμός θα έχει ε, μεγαλύτερες εξουσίε ε, όσον αφορά την έρευνα και τα πιλωτικά προγράμματα. Προβλέπει επίση η πρόταση την ύπαρξη ενό μηχανισμού ελέγχου των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θα εξασφαλίζει ότι ανακριβή και ε, ασυνεπή δεδομένα θα εντοπίζονται αμέσως. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και έχει αποτελέσει πρόβλημα γιατί τα κράτη-μέλη πολλές φορές δεν είχαν στείλει ακριβή ε, δεδομένα ε, ούτε συνεπή και πρέπει να καλύψουμε τι βάσει δεδομένων. Όσον αφορά τη διαλειτουργική ε, η πρόταση αφορά την ανάπτυξη των κυρίων ε, τεχνικών χαρακτηριστικών ε, της προσέγγισης Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν κάποιε πτυχές όμως ε, της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων ε, και βελτιώσεων κατά την άποψή μου. Το αναφέρω αυτό στην έκθεσή μου και θα το αναφέρω και σήμερα. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα της αρρωγής προς τα κράτη-μέλη. Η ικανότητα της υπηρεσίας να παρέχει αρρωγή στα κράτη-μέλη αν το ζητήσουν η ζητημάτων ε, είναι ένα από, τα, από τις πιο ε, σημαντικές αλλαγές ε, στη νέα εντολή του οργανισμού. Μιλάμε για νέα συστήματα πληροφορικής και βεβαίως τα κράτη-μέλη θα έχουν ερωτήσεις και θα ζητήσουν διευκρινήσεις, οπότε θα απευθυνθούν στο EU Στο άρθρο 12 εγώ προτείνω η τρέχουσα πρακτική για την υποβολή αιτήματο ε, στην υπηρεσία από ένα κράτος μέλος ε, για να ζητήσει δηλαδή διευκρινήσεις θα έπρεπε να πηγαίνει απευθείας ε, στην υπηρεσία και να μην περνά μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως συνέβαινε στο παρελθόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει έναν εκ έναν, έναν εκ προτέρων έλεγχο έλεγχο και θα υπάρχει και διαβούλευση πρέπει να απαντήσει επίσης εγκαίρως τα κράτη-μέλη στα, τα οποία έχουν θέσει τα ερωτήματα. Δεύτερο ε, σημείο ε, επί του οποίου ζητώ αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές εγκαταστάσεις πιστεύω ότι πρέπει η υπηρεσία να μπορεί να αντιδρά ταχύτατα ε, και να μπορούμε δηλαδή να εφαρμόζουμε νέες νομοθετικές προτάσεις μελλοντικές υπό τα υφιστάμενα τεχνικά μέσα. Συνεπώς πρέπει ε, να βελτιωθεί και ο ιστότοπος της, ε, του υπηρεσίας γιατί είναι γνωστό ότι οι νέες βάσεις δεδομένων δημιουργούνται συνεχώς. Οποιασδήποτε δηλαδή δυσκολίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει ε, τώρα ε, το νέο ε, σύστημα θα αποθηκεύεται ούτως ή άλλως, ε, τα, τα στοιχεία θα αποθηκεύονται ούτως ή άλλως στο Στρασβούργο που βρίσκονται οι βασικές εγκαταστάσεις ε, του EU Θα ήθελα λοιπόν αλλαγή στο άρθρο 13 ε, για τη δημιουργία κι άλλων τεχνικών εγκαταστάσεων αν χρειάζεται κατόπιν του Διοικητικού Συμβουλίου του EU και κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε λοιπόν ε, η κύρια εγκατάσταση βρίσκεται στο Στρασβούργο, εκεί αποθηκεύονται τα περισσότερα δεδομένα και να υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις σε άλλες ε, σε άλλες ε, περιοχές αν χρειαστεί ή αν καταστεί αναγκαίο μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τώρα το εφεδρικό σύστημα, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο και η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτρο... με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να μπορεί να αποφασίσει κατά πού θα έπρεπε να υπάρχει ε, αυτή η εφεδρική εγκατάσταση για να εξασφαλίζεται η ε, λειτουργία του συστήματος. Επίσης πιστεύω και το τόνισα ότι το εφεδρικό ε, σύστημα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει τη λειτουργία και στην περίπτωση ε, που ε, δεν λειτουργεί οποιοδήποτε σύστημα. Δεν έχω πολλά ακόμη να πω. Η συμμετοχή των ε, χωρών ε, και των χωρών που συνδέονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν ε, και των μέτρων των σχετικών με το Eurodac. Το ανέφερα σε σχέση με το άρθρο 38 ε, εγώ θα ήθελα να διευρύνω την συμμετοχή και άλλων χωρών ε, σε οποιαδήποτε άλλη ε, συμφωνία διευκόλυνσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γεωργία και Ουκρανία για παράδειγμα. Μία νέα πρόταση επίσης για ένα νέο άρθρο 38α για να υπάρξει επαρκής νομική βάση ε, για τον οργανισμό, ώστε μετά από διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να διατηρεί ε, τις σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς. Τώρα, η αποζημίωση, αλλαγές στο άρθρο 37 προβλέπει τη νομική βάση για τη συνεργασία με τους, ε, τα όργανα και τους φορείς και τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση οι υπηρεσίες που παρέχονται από το EU Lisa μπορεί να έχουν έναν αντίκτυπο στον ε, ε, προπολογισμό του οργανισμού και συνεπώς πρέπει να υπάρχει μια κάλυψη. Ένα ακόμη σημείο για τη διαφάνεια. Έχω υποβάλει τροπολογίες για την αύξηση της διαφάνειας του EU Lisa και σε σχέση με την πρόληψη της ε, σύγκρουσης συμφερόντων του Διοικητικού Συμβουλίου του εκτελεστικού διευθυντή και των μελών των ε, συμβουλευτικών ομάδων του Ήγιου Και θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι ο διευθυντή πρέπει να είναι ανεξάρτητο και δεν θα ζητήσει οδηγίε ε, από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τώρα, η εντολή του διευθυντή αυτού, εγώ προτείνω να ευθυγραμμιστεί ε, με την πρόταση για την διεύρυνση του εκτελεστικού διευθυντή, όπως γίνεται και για την Europol, δηλαδή να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα ε, διεύρυνσης ε, της θητείας μέχρι τα πέντε έτη. γιατί έχει ξανασυμβεί αυτό υπό το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο. Μία μεταβατική περίοδος δηλαδή μεταξύ του τρέχοντος νομοθετικού πλαίσιου και του επομένου. Εν κατακλείδη λοιπόν έχω καλύψει πιστεύω τα σημαντικότερα ζητήματα και θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει μία πρόκληση σήμερα να παραμείνει ανοιχτή αλλά να παραμείνει και ασφαλής. Οπότε ο ίδιου Λίσα χρειάζεται μία ισχυρότερη εντολή και επαρκή ευελιξία προκειμένου να επιτύχει αυτό το στόχο, να παραμείνει ανοιχτή αλλά να παραμείνει και ασφαλής. Με χαρά λοιπόν θα περιμένω τις απόψεις των συναδέλφων και ελπίζω να φτάσουμε σε συμφωνία σύντομα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές για το ΕΛΚ. Η Μπάρμπαρα Κουκίτσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο ε, έκθεσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ενίσχυση του οργανισμού, κάτι το οποίο συνάδει με τις προτεραιότητες του ΕΛΚ. Επίσης χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που βλέπω μια δυνατότητα περαιτέρω τεχνικών εγκαταστάσεων, την επανεισαγωγή της διάταξης που αφορά την ανεξαρτησία του εκτελεστικού διευθυντή, όπως επίσης και την ενίσχυση του άρθρου 38 παράγραφος 1 όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών που έχουν ε, συνδεθεί μέσω διαφόρων συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επιπλέον όμως ε, τροπολογίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να εξαιτιαστούν σε σχέση με το εξειδικευμένο προσωπικό, τις ανάγκες πριν από τη δημιουργία επιπρόσθετων τεχνικών εγκαταστάσεων, αλλαγές στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στη λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση του οργανισμού και ευθυγράμμιση με το πακέτο αναδιατύπωσης του SAS. Λοιπόν, θα υποβάλω ούτω ή άλλω αυτέ τι τροπολογίε σε σχέση με τα ε, σημεία αυτά. Όπω είπα και την περασμένη φορά, το EU LISA είναι μια τεράστια πρόκληση. Έχει να αντιμετωπίσει τεράστια πρόκληση λόγω των νέων τη καθηκόντων. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσει σωστά κατά τα επόμενα έτη. Αναμένω εναγωνίω στη συμμετοχή με του υπόλοιπου σκιώδει συζητητέ επί του θέματο αυτού. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσινίτσι. Ε, <clears throat> Στο Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβέη που παρουσίασε την έκθεσή της για τη νέα πρόταση καονισμού για την Ιουλίζα που θέτει τις βάσεις για έναν επικοδομητικό διάλογο ε, για να προετοιμαστεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τροποποίηση του καονισμού είναι πάρα πολύ σημαντική, ε, δεδομένου του ρόλου που θα παίξει η Ιουλίζα σε διάφορα πεδία που Παιδί που αφορούν πάντα την ανταλλαγή πληροφοριών και την ασφάλεια. Ανάλυσα με προσοχή την αρχική πρόταση τη Κομισιόν και την έκθεση τη συναδέλφου τη κυρία Μακοβέη και θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία επί των οποίων μαζί με του άλλου κοιόδη συζητητέ θα πρέπει να προβληματιστούμε. Καταρχά, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να αναλύσουμε το ρόλο τη εποπτεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη δραστηριότητα τη ε, η η τροποποίηση της εισηγήτριας ε, είναι γενικά θετική, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ε, σωστής και ελέγχου και την ε, βασική ε, ελευθερία δράσης που θα δώσει τότε στην Ιουλίζα να παίξει πραγματικά με αποτελεσματικότητα το ρόλο της. Ε, ε, κάτι άλλο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ο μηχανισμός ε, οικονομικής αντιστάθμισης που προτείνει η συγγήτρια. Νομίζω ότι και από αυτού θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ για να μην να ε, κινδυνέψουμε η υπηρεσία αυτή, ο οργανισμός αυτός να θεωρηθεί σε ένα είδος πάροχος υπηρεσιών για τον οποίο πληρώνουμε και από πάνω. Θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα κάποιοι δημόσιοι φορείς να αναπτύσσουν και να θέτουν στο εμπόριο κάποια προϊόντα σε ένα περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά μπορεί να έχει και αρνητικέ επιπτώσει, μπορεί να δημιουργήσει επικρίσει, μπορεί επίση να έχει και επιπτώσει αρνητικέ στι επιδόσει του οργανισμού, του Ιουλίζα. Ένα άλλο σημείο επίση που θα πρέπει να μα απασχολήσει περαιτέρω είναι οι συμφωνίε με άλλε διεθνεί οργανώσει. Νομίζω ότι για τη νέα παράγραφο του άρθρου 38 θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καλύτερα το πνεύμα το οποίο οδήγησε σε αυτή την αλλαγή που προτείνει η εισηγήτρια. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες για, την, για διορισμό του Γενικού Διευθυντή, οι διαδικασίες θα πρέπει να θυγραμμιστούν με τον άλλων υπηρεσιών στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων ε, και να προβλέψουμε έναν βασικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ένας από τους ε, συνομοθέτες με το πιο σημαντικό καθήκον εποπτείας του οργανισμού Ιουλίζα που θα πρέπει να το δούμε να υλοποιείται τα επόμενα χρόνια. Ε, τώρα, για τη διαλειτουργικότητα, άρθρο 9 της ε, αρχικής πρότασης της Κομισιόν, θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με τη γενική θέση, ότι αυτό το καθήκον του, της Γιουλίζα να αναπτύξει τέτοια συστήματα υπάρχει μόνο αν το αποφασίσουν οι συνομοθέτες μέσω των κατάλληλων νομοθετικών ε, κειμένων που αυτή τη στιγμή σε φάση διαπραγμάτευση. Επίσης είναι λογικό να παίξει ο, ο Ιουλίζα ε, να εξασφαλίσει ας πούμε, την διαλειτουργικότητα λόγω της επαγγελματικότητα που έχει ο οργανισμός. Κάτι που πρέπει να σας απασχολήσει περαιτέρω είναι ε, αυτό που είπε ο Ευρωπαίος Επόπτης για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ε, στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα που, δημιου... που ανέφερε ο Ευρωπαίος Επόπτης. Ε, ε, χρήση ανώνυμων στοιχείων ε, για συντηρητικούς λόγους. Ε, επίσης, τα στοιχεία του άρθρου 12.2, το οποίο έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική δομή των συστημάτων πληροφορικής. Πιστεύω ότι θα έχουμε σίγουρα την δυνατότητα συναντήσει με τους Σάντου, τους και όλους να εμβαθύνουμε στα σημεία που σας ανέφερα Και είμαι πεπισμένη ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό κείμενο που θα μας βρίσκει όλους σύμφωνους, γιατί ο σημαντικός ρόλος της ε, Ιουλίζα δεν αμφισβητείται και άρα θα πρέπει να δούμε όλο αυτό το θέμα με τεράστια προσοχή και ζήλο. Δεν υπάρχει άλλος και ο συζητητής. υπάρχει κάποιος άλλος βουλευτής που θέλει να πάρει το λόγο. Ε, το είπατε και εσείς ότι και εγώ είμαι σκιώδης συζητητής. Νομίζω ότι οι τρεις που μιλήσατε αναφερθήκατε στα πιο σημαντικά σημεία. Επομένως, περιμένω να ολοκληρώσουμε και εμείς τη δουλειά για το φάκελο αυτό. Η υποστήριξη για αυτόν τον οργανισμό είναι σαφής. Και το θέμα είναι ποιες ασφαλιστικές δικλείδες θα δημιουργήσουμε, ούτως ώστε να τηρήσουμε και τα πρότυπα τα οποία έχουμε θέσει. Κυρία Μακοβέη, για να απαντήσει. Και αν μου επιτρέψετε να δώσω και το λόγο στην Κομισιόν για να, πάρει, να πει δυο λόγια σύντομα πριν να δώσω το λόγο στην κυρία Μακοβέη. Κύριε Μίλο, πολύ γρήγορα να μας πείτε τον, την άποψή σας. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης για την πρόταση Γιουλίζα. Η Επιτροπή δέχεται μία σειρά από τις ε, ε, προτινόμενες τροπολογίες, καθώς ε, προσθέτονται νέα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα. Ωστόσο, μας προγραμματίζουν ορισμένες από τις τροπολογίες. Θα θέλαμε να σταθούμε πρώτα στην τροπολογία 1, 18 και 19 σχετικά με το άρθρο 13 που αφορά περαιτέρω ε, τεχνικές ε, προδιαγραφές που μπορούν να θεσπιστούν μετά την, ε, τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήδη προκύπτει από την αρχική πρόταση που δεν είχε υιοθετήσει η Επιτροπή τότε, γιατί ε, τα συστήματα και η τοποθέτησή τους προβλέπεται στα ίδια τα συστήματα υπό τον κανονισμό VIS, SIS. Που αναφέρεται ξεκάθαρα τοποθεσία. Οποιαδήποτε λοιπόν αλλαγή στην τοποθεσία ε, απαιτεί αλλαγή και των μέσων αυτών. Και κατά τη γνώμη μας αυτό δεν είναι απόφαση που μπορεί να πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το κείμενο έχει τροποποιηθεί για να επιτρέπει τη λειτουργία, ταυτόχρονα λειτουργία των ε, εφεδρικών ε, συστημάτων. Είναι κάτι το οποίο έχει ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Εμείς θεωρούμε ότι είναι ε, επιλεγεί το active-active. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με την τροπολογία 18 στη διατύπωση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε επίση και με τα 19 που προβλέπει ότι ε, η εφηδική τοποθέτηση θα θεσπιστεί βάσει οποιασδήποτε άλλη απόφαση ε, του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι η τοποθεσία του εφεδρικού συστήματος μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια κατόπιν απόφαση του Συμβουλίου. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει εξολόγηση αντικτύπου που να δεκμηριώνει την ανάγκη τέταρτης τοποθεσίας ή μεταφοράς του εφεδρικού συστήματος. Υπάρχει λοιπόν η ευελιξία χρήσης ε, του εφεδρικού συστήματος ως ε, μη ενεργού και αυτό ήταν και μία από τις επιλογές που είχε παρουσιάσει ο τελευταίος Διευθυντής στο Συμβούλιο σε 9 Οκτωβρίου και νομίζω ότι αυτό ναι, θα πρέπει να διατηρηθεί ως τεχνική λύση. Κλείνοντας, όποιες αποφάσεις έχουν να κάνουν με αλλαγές στην, στην νομοθεσία πρέπει να αποφασιστεί από τους νομοθέτες ε, βάσει μιας αξιολόγησης αντικτύπου και αυτό δεν είναι αποφάση που μπορεί να πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 3 και 16 που σχετίζονται με το 12α, στήριξη προς ε, κράτη-μέλη μπορεί να διευκρινιστεί η διατύπωση, δηλαδή ότι αυτέ οι νομοδοτήσει θα πρέπει να υποβάλλονται απευθεία στον οργανισμό. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το αίτημα επιπλέον ε, στήριξη που απαιτείται σε περίπτωση έκτακτων μέτρων σχέση με την ασφάλεια ή τη μετανάστευση, αυτά θα πρέπει να απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είναι η Επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να αξιολογήσει την ασφάλεια ή τις μεταναστευτικές ανάγκες. Αυτή τη διαδικασία ακολουθήσαμε στις αρχές του 2016 όταν η Επιτροπή προσκάλεσε την Ιουλίσσα να παρέχει στήριξη στα hot spots ε, εν μέσω της προσφυγικής κρίσης. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι να προσθέσουμε ότι θα προχωρήσουμε κατά πόσο υπήρξε έγκαιρη απάντηση από πλευρά του οργανισμού προ τα αιτήματα των κρατών Για την τροπολογία 4 και 17. Διακόπτει ο πρόεδρο, Συγγνώμη, αλλά σε δύο-τρία λεπτά πρέπει να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Είναι και μακροσκελής. Μπορείτε να ολοκληρώσετε παρακαλώ και τις ειδικέ συστάσεις για τις τροπολογίες μπορείτε να τις στείλετε και γραπτός ε, στην εισηγήτρια στη συνέχεια. Μάλιστα. Προτείνω να συναντηθούμε με εισηγητικές και όδους εισηγητές για να εξετάσουμε ακριβώς τις τροπολογίες. Okay, thank you very much for, for that uh, understanding. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε για την κατανόηση. τα σημειώνουμε όλα αυτά. Να δώσουμε και πάλι το λόγο τώρα στην εισηγήτρια, κυρία Μακοβέη, πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι έχουμε και άλλη ψηφοφορία για την προστασία δεδομένων. Υπήρξε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πριν από καιρό όταν ε, συστάθηκε η Γιουλίσσα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι πιο ασφαλές ένας οργανισμός να αναλάβει όλες αυτές τις φάσεις δεδομένων από πλευράς ε, προστασίας δεδομένων και ουδετερότητας. Και όλοι ξέρουμε ότι ε, το προσωπικό του Λίσσα e δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των βάσεων δεδομένων των εξυπηρετητών. Πάντα λοιπόν είναι πιο εύκολο να έχουμε έναν οργανισμό για την βάση δεδομένων από ότι 10 για την προστασία δεδομένων από ότι να έχουμε 10 ξεχωριστές υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε. Να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι ε, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 6 Νοεμβρίου, 6 Νοεμβρίου, 6 το απόγευμα. Θέλουμε εδώ λοιπόν αυτό το σημείο να αφήσουμε ένα λεπτό στους συναδέλφους για να καθίσουν πριν ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία.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 Colleagues, Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. I παρακαλώ και τελευταίοι. Πρώτη η ηλεκτρονική ψηφοφορία της δεύτερης φουρνιάς για την ε, στρατηγική, την ψηφιακή. Αντζέλικα, θα πάρεις το λόγο. Συμβαστική 3. Έναρξη. Συνεχίζει την ψηφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 26. Άρχεται. Απορρίπτεται. Σεβαστική 4 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνομαστική 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. συμβαστική. Άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται τριάντα εφτά πρώτο τμήμα άρχεται πέρας απορρίπτεται σαράντα τρία τροπολογία άρχεται Πέρασε. Ένας παραπάνω τους σοσιαλιστές εδώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Ετολογικέ σκέψεις, τροπολογία 7, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Πέρας. Και πάλι ένας παραπάνω από τους σχελιστές. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ, βγάλτε μια κάρτα. Ευχαριστώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Έναρξη. Πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 έρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 15. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 16. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 17. Έναρξη. Πέρας. Εκκρίνεται. Συμβαστική 1. Έναρξη. Πέρας. Έγινε ανατά. Τροπολογία 22. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρασε. Έγκρινεται. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. Επί του κειμένου όσο έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έγκρινεται. 52 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Στην κυρία Μιλνάρ. Colleagues, Στην έκθεση για το σεβασμό της ιδιωτική σφαίρα και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές Κατάσταση Κατάρτιση οδηγία 2002 58 ΕΚ, κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η εισηγήτρια κυρία Μάριου Λόριστην. Υιοθέτηση του σχεδίου έκθεσης. Θέλει να πάρει το λόγο η συγγήτρια πριν πάμε στην ε, ψηφοφορία. Μάριου, σύντομα. Να ευχαριστήσω όλους τους και συγγητές και του ΕΛΚ που κάνανε προσπάθειες μέχρι τελευταία στιγμή για να πετύχουμε τους συμβασμούς. Δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όλα κατευχήν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, ε, τεράστια πίεση και ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην ομάδα. Για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Φτάσαμε όντως στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ξεκινάμε τον συμβασμό άρθρο 1. Συμβασμό για το άρθρο 1. Ψηφίσουμε τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα παραπάνω. Ένα βουλευτή παραπάνω, παρακαλώ, κανονίστε. Εντάξει. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 2. Συμβασμός για το άρθρο 2. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 3. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 4. Ψηφίσουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 5. Ψηφίσουμε τώρα, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 6. Ψηφίζουμε τώρα παρακαλώ. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 7. Ψηφίζουμε τώρα. την ησυχία σας. Δεν θα σας, δώσω, δεν θα σας πω τους αριθμούς των σελίδων. Συμβιβασμό επί του άρθρου 7. Βρείτε τον με την ησυχία σας. Κυρία Στίβενς. Το βρήκατε, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό για, για το άρθρο 8. Ψηφίζουμε. Όσο και να με ρωτάτε, δεν σας, θα σας πω τον αριθμό των σελίδων. Μπορείτε ακόμα να ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 9. Ψηφίζετε τώρα. Εγώ θα περιμένω μέχρι να ψηφίσουν όλοι. Συμβασμός για το άρθρο 9. Ακόμα μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας φοφορίας Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 10. Ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Ακόμα μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 11α. αέρας προφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στο συμβασμό για το άρθρο 12. Όχι, δεν θα ψηφίσουμε τα άλλα, γιατί ο συμβασμός για το 11α υιοθετήθηκε. Πάμε λοιπόν στον συμβασμό για το άρθρο 12. Συμβιβασμός για το άρθρο 12. Ακούστε τι σας λέω. Μπορείτε ακόμα να ψηφίσετε για το συμβασμό για το άρθρο 12. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 13. Ψηφίσουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, Συμβιβασμός για το άρθρο 11, ε, 14, συγγνώμη. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας προφορία συγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 15. Πέρας Συμβασμός για το άρθρο 16. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 17. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 18. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 19. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 21. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 22. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός για το άρθρο 23. Πέρας ψηφοφορίας. Συμβασμός για το άρθρο 24. Πέρας φοφορίας, Εγκρίνεται για το άρθρο 25. Πέρας φοφορίας, Εγκρίνεται συμβασμός για το άρθρο 26. Πέρας φοφορίας, εγκρίνεται συμβασμός για το άρθρο 27. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τις αιτιολογικές σκέψεις, καλύπτονται όλες. Πάμε στο, στην ψηφοφορία του τροποποιημένου κειμένου, ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. είναι σε δύσκολη θέση. Αν η Επιτροπή συνολικά θέλει να περιμένουμε ένα λεπτό. Για την τελική ψηφοφορία δεν μιλάμε. Ναι. Μια στιγμή, συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ένα ε, συντονιστή μα ζήτησε να κρατήσουμε λιγάκι πιο ε, ανοιχτή μάλλον την ψηφοφορία για περισσότερο. Ε, κλείνει όμω τώρα, εγκρίνεται 31 υπέρ, 24 κατά, μία αποχή. Ψηφίσουμε για την εντολή για διπραγματεύσει. Ψηφίστε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Ακόμα ψηφίζετε. Λήξη. Εγκρίνεται 31 ψήφι υπέρ, 25 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Κύριε Μπόνη, θέλετε να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, συνοδεύει ο κύριος Μπόνη. Η κυρία Μάριου Λόριστον ε, περνάει τις βερθές τις μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αποφασίζει να μεταπηδήσει στην Εστονία. Θα συνεχίσει εκεί την καριέρα της. Την ευχαριστώ λοιπόν ε, πολύ για την ε, συνεισφορά της στην δύσκολη αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ Μάριου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, αξιοπρεπής παρατήρηση. Και καλή τύχη, Μάριου. Πολύ ενθουσιασμό είχατε όλη για αυτή την ψηφοφορία. Πάμε στην επόμενη όμως, σας παρακαλώ. Υπάρχουν και χρονικές πιέσεις ε, που βαραίνουν πολλούς από εμάς. Ας τους σεβαστούμε, τους αδέρφους αυτούς που πιέζονται χρονικά. Πάμε τώρα. Στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή στην Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, η συγκητή είναι ο Άξελ Βος. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές Πήγε αρκετά σύντομα, έτσι, ομαλά η συνάντηση, παρότι μας καθυστέρησε αρκετά. Ε, και το αποτέλεσμα νομίζω ότι μπορεί να μας ικανοποιήσει όλους. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Άξελ. Πάμε στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 187. Ψηφίστε τώρα. Okay. Ε, Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Λήξη προφορίας. Εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 8. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβασμός A. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός B. Πέρας. Εγκρίνεται. συμβασμό C. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Συνάδελφοι. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 14. Έκανα λάθος. Τροπολογία 14. Ψηφίσουμε τώρα. Μπορεί να ψηφίσετε ακόμα. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα τροπολογία 17. πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2.42. Ψηφίζεται. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβασμός D. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός E. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Δεξί. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός F. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός G. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός H. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβασμός I. Λήξη. εγκρίνεται. Κοντ 15. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός J. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός K. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός L. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 284. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 1. Λήξη. Γκρίνεται. Συμβασμός O. Λήξη. Γκρίνεται. Τροπολογία 69. Τροπολογία 69. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τζούρι 40. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός P. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός Q. Λέξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Λέξη. Εγκρίνεται. Τζούρι 42. Λέξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός R. Λέξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός S. Λέξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός T. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός ZD. Ο συμβασμό για την προστασία των δεδομένων. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός TA. Λέξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός U. Λέξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός B. Β, συγγνώμη. Λέξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός W. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 387. 387. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός 6. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός Y. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός Z. Λήξη. Γίνεται. Τροπολογία 142. Λήξη. Εγκρίνεται. 143. Τοπολογία 143. Ψηφίζουμε τώρα. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 144. Λήξη. Εγκρίνεται. 145. Ψηφίζουμε χρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται 146. Ψηφίζουμε τώρα. Λήξη. Εγκρίνεται 147. Λήξη. Εγκρίνεται 148. Λήξη. Εγκρίνεται. 149 και κοντ 43 μαζί. Λήξη. Εγκρίνεται. 150. έκπληξη. Εγκρίνεται. 151 έως 154 μαζί. Ένα ψηφοφορίας. Λήξη. Γκρίνεται 155. έκπληξη. Κοντ 44. Λήξη. Απορρίπτεται. Κοντ 45. Ψηφίζουμε τώρα. Λήξη. Πέρασε. Απορρίπτεται. 156. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 175. Πέρας. Εγκρίνεται. 158. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. 408 και Λάθος, λάθος, συγγνώμη. 408. Πέρας. Απορρίπτεται. 159 τώρα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Κον 46. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 160. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 409. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Κοντ 48, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Κρίνεται. Κοντ 48, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ζήτα σι άρχεται. closed. Πέρας. Συγγνώμη συναδελφοί, κάτι έγινε με τα μηχανήματα ψηφοφορία. Λοιπόν, να ξανακάνουμε τη συμβαστική ZC. Γιατί δεν γράφτηκε στο μηχάνημα. Λοιπόν, ξανααρχίζει η ψηφοφορία. ZC. ZC. Άρχεται. ZC. Συμβιβαστική. Ζήτα Σι παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τζούρι 52. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 165. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 166 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 167 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 168 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 169. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Κοντ 50 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 170 άρχεται. Και κον 51. 170 και κοντ 51 από εκείνου άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Κόν 52 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 171 και κοντ 53 μαζί άρχεται. Πέρασε. Πέ, ε, πέρασε μάλιστα. Δεκτή. Κοντ 54 άρχεται. Πέρασε. Δεκτή. 172 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 173 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 174 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 4.73. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 4.14. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 175. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τσούρι 58 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 176 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 177 άρχεται. Πέρας. Ναι. Απορρίπτεται. 178 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 179 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 180 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 181. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 4-16. Ε, Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τζούρι 61. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 182 και 417. Από κοινού άρχεται. Πέρας. Δεκτές. 418 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 183 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 184 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 185 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 186. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Κοντ 55. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Κοντ 56. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αν αιτιολογικές σκέψεις και αναφορές 188 και 189 από κοινού. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τζούρι. Α, όχι. Όχι. Συμβαστική α, άρχεται. Ζ κεφαλαίο α μικρό άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τζούρι 2 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τζούρι 3 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τζούρι 4 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τζούρι 5 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τζούρι 7 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 198 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 199 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Κοντ 3 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τζούρι 8 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τζούρι 9 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 201 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική ZB άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2.13 άρχεται. 2.13. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 5 και τζούρι 14 μαζί. 5 και τζούρι 14. Πέρας. Εγκρίνονται. 2-15. άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τζούρι 15, άρχεται. Πέρασε. Δεκτή. 2-16, άρχεται. Πέρασε. Δεκτή. 2-17, άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Κοντ 5. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Κοντ 6. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τζούρι 16. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 2.18 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.19 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 2.20 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τώρα να ψηφίσουμε το κείμενο ως τροποποιήθηκε ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, 0 αποχές. Και τώρα να ψηφίσουμε για την απόφαση να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 50 υπέρ, 5 κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. colleagues, um, colleagues, just uh, for your timings and information. Συνάδελφοι, τελειώσαμε νωρίς την ψηφοφορία, οπότε θα κάνουμε διάλειμμα μέχρι το επόμενο θέμα, που θα είναι στις 12.30, γιατί θα κάνουμε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε συνεχίζουμε στις 12.30 για με την κοινή συνεδρίαση με την Οικονομική Επιτροπή. Άρα, διακοπή και διάλειμμα μέχρι το 10.30. Και σα ευχαριστώ για τις συνεργασία σα όσον αφορά τι ψηφοφορίε πέρα ψηφοφοριών. Ξαναρχίζουμε στο δεκάμιση.